Bien. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons. Euh, ε, κυρίε και κύριοι, θα αρχίσουμε. Η κατάσταση σήμερα είναι κάπω χαόδη όσον αφορά την κυκλοφορία στου δρόμου. Δείξτε σα παρακαλώ κατανέωση για του συναδέλφου που ήταν καθυστερημένοι. Ζητούμε συγγνώμη για την κάποια καθυστέρηση. Αλλά καλό είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά. Γιατί οπωσδήποτε οι συνάδελφοι που λείπουν θα έρθουν. Με κάθε Η συνεδρίασή σήμερα είναι δημόσια ακρόαση για το θέμα των, ε, της άμυνας κατά των ε, ρουστικών πυράβλων. Ξέρετε, είναι σημαντικό γιατί με διάσκεψη κορυφή τη Λισαβόνη τη περασμένη εβδομάδα ένα από τα κύρια αποτελέσματα που τονίστηκαν στη εθέτηση μιας νέας στρατηγικής ε, αντιμετώπισης αφορά ακριβώς το δυναμικό που πρέπει να αποκτήσει το ΝΑΤΟ στον τομέα των βαλιστικών πυράβλων για να μπορέσει να προστατεύσει τους ε, λαούς και τους χώρες της συμμαχίας. Διαφέρει το σημερινό πρόγραμμα που υπάρχει για την πολυμερή ε, άμυνα που καλύπτει τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Το θέμα αυτό είναι ελευ... Ε, ευαίσθητο συγγνώμη, πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Στο επίκεντρο της ε, συμμαχίας, εκείνους που θεωρούν το δυναμικό αυτό είναι συμπληρωματικό της ε, πυρηνικής ε, απόκρουσης, άλλοι θέλουν να είναι ε, υποκατάστατο. Υπάρχει συζήτηση και με τους εταίρους της συμμαχίας, Ρωσία κυρίως, και στο εσωτερικό της συμμαχίας, για να ανοιχτευτούν οι απειλές που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την ανάπτυξη του προγράμματος αυτού. Έχουμε ένα κείμενο επιτάκτος και η απόφαση σημειώθηκε όπως ε, μας το είπε και ο στρατηγός Μπριάλ που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο για την καλή οργάνωση της ακρόασης. Έχω να σας πω ότι έχουμε τέσσερα πάνελ Κάθε παρουσιαστή θα έχει περίπου 10 λεπτά για την εισαγωγική του παρουσίαση και μετά θα πάει ζήτηση. Η πρώτη θα γίνει με τον κύριο Περ που εκπροσωπεί το Υπουργείο Άμυνες των Αμερικής και θα μας παρουσιάσει βέβαια την άποψη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Το δεύτερο πάνελ θα υποδεχθεί τον πρέσβη της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρογκοζίν που είναι εδώ μαζί μας. Το τρίτο πάνελ θα έχουμε τον κύριο Ζάντρα από τον ΝΑΤΟ και τον Καμίλ Γκρό από το Ίδρυμα για τη Στρατηγική Άμυνα του Παρισίων και το τελευταίο πάνελ θα έχει σαν στόχο την βιομηχανική πτυχή. Θα μας μιλήσει η κυρία Βερονίξα Μελάκ και ο στρατηγός Μπερνάρ Λιμπά, που είναι σύμβουλος Δύο επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί στο πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, μια που έχουμε ήδη κάποια καθυστέρηση, δεν θέλω να αναπτύξω ιδιαίτερα το θέμα της εισαγωγή. Θα έρθω να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέλ και μετά την παρέμβασή του θα συζητήσουμε του θέματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εμείς ε, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό για να σας δώσουμε κάποιες ε, πληροφορίες. Βλέπω πως δεν υπάρχει μετάφραση από τα δανέζικα, άρα λοιπόν ίσως καλύτερα θα ήταν να μιλήσουμε αγγλικά σήμερα το πρωί. Να σας πω πως είναι ιδιαίτερα τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ ε, σήμερα το πρωί. Έχουμε εδώ τον κύριο Ρογκόζιν και πολλούς ομιλητές, όπως επίσης και τους αξιότιμους ευρωβουλευτές. Και η ευκαιρία που μας δίνει αυτή η δημόσια ακρόαση είναι μια την οποία χαιρετίζουμε ιδιαίτερα και νομίζω ότι ε, ήταν μια εξαιρετική σκέψη να μας υποδεχθείτε εδώ και μάλιστα σας ε, συγχαίρω που με τέτοιο καιρό καταφέρατε να φτάσετε. Πρέπει να σας πω πως για 18 χρόνια εγώ ε, ήμουν το Κογκρέσο, ε, εργαζόμουν εκεί και σε 12 και 12 χρόνια ήμουνα σε επιτροπές της Γερουσίας που ε, ήταν αρμόδιες για τέτοιου είδους θέματα. Καταλαβαίνω λοιπόν πως και η δική σας επιτροπή ε, έχει ως βασικό στόχο να κατανοήσει το ευρύ κοινό τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο αυτό της άμυνας και είναι πολύ σημαντικό το κοινό να δείξει κάποια κατανόηση για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και για τα όσα ε, θα κάνουν από κοινού το ΝΑΤΟ και η Ρωσία και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι κοινέ τους προσπάθειες θα επηρεάσουν την Ευρώπη. Ε, ξέρω πως εσείς έχετε επιπλέον αρμοδιότητες εδώ στο Κοινοβούλιο από τότε που ετέθησε ισχύ η ε, συνθήκη της Λισαβόνες και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά στο νέο πλαίσιο των αμυντικών προσπαθειών στην Ευρώπη. Η Λισαβόνα είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία και πρέπει να σας πω πως ε, ήταν σημαντικό για μας να βρεθούμε σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο πριν από 10 μέρες για την σύνοδο που έγινε εκεί το περασμένο Σαββατοκύριακο πιο συγκεκριμένα. Και δεν θα πω σύνοδο, θα πω για τι συνόδου στον πληθυντικό, γιατί παράλληλα στι δύο ημέρε που ήμασταν εκεί έτρεξαν τέσσερι σύνοδοι. Είχαμε ε, του 49 αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων ε, που συμμετέχουν στι επιχειρήσει του Αφγανιστάν. Είχαμε τη σύνοδο. Ε, μεταξύ του Προέδρου κ. Ομπάμα και της ηγεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με τα μέλη της Συμμαχίας, και βεβαίως το Συμβούλιο σε επίπεδο αρχηγών ε, ε, κρατών μεταξύ ε, ΝΑΤΟ και Ρωσίας όπου όλοι οι αρχηγοί κάθισαν σε ένα τραπέζι και έλαβαν αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο 29 μελών. Πρέπει να σας πω πως Είχαμε λοιπόν τη σύνοδο της συμμαχίας και τις συζητήσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και θα σας δώσω όσες πληροφορίες θέλετε και μετά θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας, γιατί από την Ουάσιγκτον αυτή είναι η εμπειρία μου ότι πιο πολύ θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις παρά να ακούσετε τη δική μου παρουσίαση. Βεβαίω, ε, το κεντρικό σημείο της ε, Συνόδου της Συμμαχίας ήταν το νέο στρατηγικό δόγμα το οποίο αποφασίσετε εκεί. Είναι ως ε, είναι το ίδιο με το επιχειρησιακό ή επιχειρηματικό δόγμα που ακολουθεί μια επιχείρηση. Είναι ένας οδικός χάρτης για το πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και πώς πιστεύουμε ποια θέματα θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες τα επόμενα δέκα χρόνια. Εκεί λοιπόν ε, λάβαμε κάποιες αποφάσεις που καλύψαμε και το θέμα της αντιπυραυλικής στο στρατηγικό δόγμα που συμφωνήθηκε 19, 19 ε, Νοεμβρίου ε, στο ΝΑΤΟ για το περιβάλλον ασφάλειας όπως το περιγράφουμε ξεκινήσαμε με κάτι το οποίο είναι ε, προφανές αλλά εξαιρετικά ευχάριστο πως αυτή τη στιγμή η περιοχή, η ευρωατλαντική περιοχή είναι ειρηνική, υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα ε, συμβατικής ε, επίθεσης και αυτό αποτελεί ένα ιστορικό κριτικό σημείο στο οποίο έχουν φτάσει οι σχέσεις μας και όπου θεωρούμε πως είμαστε πολύ επιτυχημένοι σύμφωνα με τους στόχους που είχε το ΝΑΤΟ τα τελευταία 50 χρόνια τώρα για την διάδοση των πυρηνικών όπλων και για τα όπλα μαζικής καταστροφής. Πιστεύουμε πως εκεί οι απειλές για την διεθνή ευημερία και η ειρήνη έχουν αυξηθεί και πιστεύουμε πως τα επόμενα 10 χρόνια θα ε, αυξηθεί ο κίνδυνος της διασποράς των πυρηνικών σε κάποιες από τις πιο ανήσυχες περιοχές του κόσμου. Και γι' αυτό το ΝΑΤΟ αποφάσισε ε, αποφάσισε για να προστατεύσει τις περιοχές μας από ε, βαλιστικές επιθέσεις ε, να στήσει μια συλλογική αντιπυραυλική άμυνα και όλα αυτά στο πλαίσιο της απόκτησης της απαραίτητης στρατιωτικής δύναμης η οποία θα εξισορροπήσει τις άλλες ε, ε, δυνατότητες που έχουμε και που θα εξασφαλίσουν τα όσα έχουμε στο άρθρο 5 της Συμφωνίας της Συμμαχίας. Είπαμε πως για την πυραυλική αντιπυραυλική άμυνα θα επιδιώξουμε τη συμφωνία με τη Ρωσία και με τους υπόλοιπους εταίρους. Στη Σύνοδο συμφωνήσαμε επίσης το ποια θα είναι η αποστολή μας τα επόμενα δέκα χρόνια. Μία δήλωση αποστολής, ένα mission ε, statement και το ανακοινοθέν, ε, το οποίο πάντα εκδίδεται μετά από τέτοιου είδες συνόδους, δώσαμε κάποιες λεπτομέρειες για τα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν τμήμα της απόφασης για την αντιπυραυλική άμυνα. Γιατί βεβαίως αυτό αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης απόκρισης κατά της διασποράς, όπως σας είπα ένα κίνδυνος ο οποίος είναι κατά τη γνώμη μας όλο και πιο ορατός και έχουμε σκοπό να καλύψουμε πλήρως όλους τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, επικράτειες και στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ που απειλούνται από βαλιστικές επιθέσεις. Θέλουμε λοιπόν έτσι να γίνει πιο ορατή η αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνει το ΝΑΤΟ και βεβαίως να γίνει ένας πιο ε, ίσως ισότιμος επιμερισμός του κόστους. Θα δούμε λοιπόν ε, το θέμα του κόστους, της τεχνικής βιωσιμότητας, όπως επίσης και του βαθμού επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτό λήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα θα χρησιμοποιήσουμε το τρέχον πρόγραμμα ε, το οποίο είναι ένα, ένα πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας και είναι το ALTPMD, το οποίο εμείς, παρόλο που είναι δύσκολο ακρόν χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια στο ΝΑΤΟ και θα το διευρύνουμε έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει πιο ευρείες περιοχές και πληθυσμούς, γεωγραφικά εννοώ. Και βεβαίως η Συμμαχία συμφώνησε να καλωσορίσει την συνεισφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στα βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής, τουλάχιστον σε δυνατότητες ραντάρ και ανάσχεσης, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε την προσαρμοσμένη στην Ευρώπη στρατηγική. Έτσι την έχουμε χαρακτηρίσει. Στη Σύνοδο αποφασίσαμε να αναθέσουμε στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ να ε, στήσει τις απαραίτητες δομές χειρισμού ε, και διοίκησης που ελπίζουμε θα εγκριθεί το Μάρτιο από τους Υπουργούς Αμήνης και να μας παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για να γίνουν όλες οι προσπάθειες, όλες οι συμβατικές ε, ε, εργασίες που θα μας επιτρέψουν να διευρύνουμε αυτή την αντιαεροπορική αντιπυραυλική άμυνα έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι μέχρι τον Ιούνιο που θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί φέτος. Όπως είπα λοιπόν και προηγουμένως, το βασικό που προσφέρει σε ραντάρ και δυνατότητες ανάσχεσης είναι υλικό το οποίο θα δώσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και το σύστημα αυτό Θα χρησιμοποιήσει και θα αναπτύξει το σύστημα αυτό σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη βασίζεται σε κρούζερ και ε, καταδιοκτικά, με συγχωρείτε, ε, ε, τον είπα, τα Aegis, τα οποία έχουν τέτοιες δυνατότητες ανάσχεσης στο σύστημα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μικρής και μέσης εμβέλειας βαλιστικών πυράβλων. Και όλα αυτά μέχρι το Δεκέμβριο του 2011. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ξεκινώντας από το 2015, αυτό το δυναμικό θα ενισχυθεί πρώτον με δυνατότητες ανάσχεσης πιο δυναμικές στα ίδια τα σκάφη και δεύτερον με την χρήση τους, ε, με την εγκατάστασή τους ε, ε, χερσαία στη Ρουμανία για παράδειγμα και το 2018 θα καλύψουμε ε, και τους βαλιστικούς πυράβλους μέσω και ε, μεγαλύτερου βεληνικούς με το δεύτερο στρατόπεδο εγκατάσταση στην Πολωνία με την δημιουργία μιας έκδοσης ε, μιας εκδοχής πιο ε, ισχυρής των βλημάτων SM3. Θα έχουμε το μπλοκ 2B που θα μας δώσουν τη δυνατότητα ή τουλάχιστον θα μας δώσουν την περιορισμένη δυνατότητα αναλόγων και με τον το αριθμό που θα αναπτυχθούν ε, βλημάτων διπυρωτικού βεληνικού, ε, που θα μπορούν για παράδειγμα ε, να απειλήσουν τις Ηνωμένε Πολιτείες από την Μέση Ανατολή, επεκτόξευση στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε λοιπόν πως το σύστημα μας είναι εξαιρετικά εξαιρετικά ευέλικτο και έχει ως σκοπό να προσαρμοστεί έτσι ώστε με ε, ε, συνδυασμό ε, αισθητήρων και ραντάρ να αντιμετωπίσουν τις απειλές αυτές, τις βαλιστικές απειλές από όπου και να προέρχονται. Και κάτι ακόμα που θα ήθελα να τονίσω πριν συζητήσουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία είναι πως για χειρισμό και διοίκηση αυτού του νέου συστήματος του ΝΑΤΟ αυτή η ε, ευρωπαϊκή προσαρμογή του συστήματος ε, και η κάλυψη της ευρωπαϊκής ε, επικράτειας όπως και οποιαδήποτε άλλα συστήματα τα οποία μπορούμε να, θα, τα οποία θα είναι διαλειτουργικά και θα, τα οποία θα προσφέρουν οι δικοί μας Ευρωπαίοι εταίροι, να σας πω πως αυτές οι διευθετήσεις χειρισμού και διοίκησης θα πρέπει με συνενετικό τρόπο από όλα τα 28 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να συμφωνηθούν στο Συμβούλιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Άρα λοιπόν πρέπει να σας πω πως όλα, όλα αυτά θα γίνουν σεβαστά. Και αυτά για τα ALT-BMD. Ή αλλιώς επιχειρησιακή αντιπυραυλική άμυνα. Για την προσέγγιση αυτή λοιπόν η οποία είναι προσαρμοσμένη στην Ευρώπη, να σας πω πως αυτό το οποίο οι ΕΕ θα προσφέρουν ως ε, εθνική συμμετοχή ε, είναι το να καλύψει το κόστος αυτής της συνεισφοράς, γιατί πρέπει να σας πω πως ε, στο Συμβούλιο στο Συμβούλιο των Εθνικών Διευθυντών Εξοπλισμών ε, το κόστος της επέκτασης του ALTBMD θεωρήθηκε πως ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ για 10 χρόνια και αυτό θα μοιραστεί ε, μεταξύ των κρατών μελών. Αν λοιπόν αφήσουμε, ε, χωρίσουμε το κόστος στα τρία, και δούμε ποιο ποσό αντιστοιχεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στους Ευρωπαίους και το διαιρέσουμε για τα 10 χρόνια, θα δούμε πως το κόστος της εφαρμογής του προγράμματος αυτού για το ΝΑΤΟ τελικά είναι χαμηλότερο από το κόστο της αγοράς ενός ε, αντιαρματικού οχήματος κάθε δύο χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν πως είναι ένα κόστος εξαιρετικά χαμηλό και δεν είναι ε, συγκρίσιμο με ε, το μέσο κόστος των εξοπλιστικών μας, των εθνικών εξοπλιστικών μας προγραμμάτων συζητήσαμε πολλά θέματα ε, και με τους Ρώσους συναδέλφους στη Σύνοδο με τη Ρωσία. Ε, χαρήκαμε πολύ που συμμετείχε ο πρόεδρος της Ρωσίας και πρέπει να σας πω πως το βασικό θέμα το οποίο κάλυψε ε, όλες τις συζητήσεις που κάναμε εκεί και ο πρέσβης κύριος ε, Ροκοζίν είναι στην αίθουσα και νομίζω θα μας τα εξηγήσει αυτά αργότερα είναι πως η συνεργασία μας ήταν εξαιρετικά παραγωγική. Οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν στη Λισαβόνα για τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Ρωσία στην αντιπυραυλική άμυνα ήταν κάποια προσωρινά συμπεράσματα, δηλαδή θα χαράξουμε ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο ακόμα δεν έχει παραδοθεί, αλλά ως συμπεράσματα ήταν πολύ βασικά. Δύο βασικές αποφάσεις πήραμε από κοινού η πρώτη σχετίζεται με την συνεργασία ε, για το TBM, βαλιστικά όπλα θεάτρου επιχειρήσεων. Εκεί θα ξανασυνεχιστεί η προσπάθεια συνεργασίας που είχε λήξει το 2008 και μέχρι τον Ιούνιο θα δώσουμε ε, σάκα και οστά σε μία συμφωνία συνεργασίας για ε, βαλιστικούς πυράβλους ε, σε ένα επόμενο βήμα παραπάνω από αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει μέχρι σήμερα και πρέπει να σας πω πως στα 29 κράτη-μέλη που συμμετέχουν ε, στο Συμβούλιο αυτό το δόγμα της ευρωπαϊκής προσέγγισης ε, στο θέμα αυτό που θα λάβει υπόψη τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας είναι η άποψη που πριτάνευσε. Πρέπει να σας πω πως δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση. Αυτό που θα λέγαμε στα αμερικανικά το ξεκινάμε από το τίποτα, δεν ισχύει. Βασιζόμαστε στα όσα έχουμε χτίσει τα πλαίσια της παλαιότερης συνεργασίας μας, γιατί μέχρι το καλοκαίρι θα συνεργαστούμε για να συμφωνήσουμε ακριβώς πώς θα ευθυγραμμίσουμε τα συστήματα της πυραυλικής μας άμυνας στα πλαίσια ενός πνεύματος σύμπνοιας και συνέργειας. Θα κάνουμε και κάποια γυμνάσια με τη βοήθεια υπολογιστή με τη Ρωσία ε, τα επόμενα 4-5 χρόνια και πρέπει να σας πω πως όταν ήμουν εγώ στο ΝΑΤΟ ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής για τους εξοπλισμούς είχα την τιμή να είμαι αρμόδιος να διαπραγματευτώ τους όρους αναφοράς για την συνεργασία αυτή με τον ε, στρατηγό Μπαγεύσκη, ο οποίος ήταν ε, ο αρχηγός επιτελείου ε, της Ρωσίας και πρέπει να σα πω πω οι διαπραγματεύσει αυτέ ήταν σοβαρέ, ήταν ενδιαφέρουσε. Τι προσέγγισαν και οι δύο πλευρέ λαμβάνοντα υπόψη τα συμφέροντά του και το γεγονό πω και οι δύο θέλουν να ορίσουν τα συμφέροντα αυτά. Και καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συνενετική απόφαση, την οποία αποδείξαμε με τα γυμνάσια και τι ασκήσει που κάναμε για διάφορα για 4-5 έτη και τον Ιανουάριο του 2008 αυτά κορυφώθηκαν με γυμνάσια που έγιναν έξω από το Μόναχο σε μια γερμανική εγκατάσταση, στρατόπεδο, που θεωρήθηκαν ιστορικής επιτυχίας. Και ξέρω πως ένας γερμανός στρατηγός είπε τότε σε κάποια συνέντευξη τύπου πως έχουμε αποδείξει πως συνεργαζόμενοι το ΝΑΤΟ και η Ρωσία χρησιμοποιώντας τους συμφωνημένους όρους ε, και δόγματα μπορεί να υπερασπιστούν οποιαδήποτε επικράτεια η περιφέρεια απειληθεί μελλοντικά. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα με τον οποίο πλησιάζουμε τη Ρωσία στα πλαίσια της αντιπυραυλικής άμυνας. Βεβαίως η Ρωσία θα δώσει μεγάλες δυνατότητες αντιβρεβλαβικές άμυνας προσφέροντας την εθνική της συμμετοχή σε αυτή τη νέα τάση συνεργασίας. Η Ρωσία ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιεί ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας ε, το οποίο καλύπτει την πρωτεύουσα Μόσχα είναι η τρίτης γενιάς αντιβαλιστική πύραυλη που είναι εξαιρετικά ε, ισχυρό αλλά λίγο περιορισμένο. Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει τη στρατηγική ισορροπία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ γιατί ε, ο αριθμός των, ε, ο αριθμός των εγκαταστάσεων ανάσχεσης που είναι εγκαταστημένα σε σιλό γύρω από την Μόσχα, σε στοές δηλαδή γύρω από τη Μόσχα, καλύπτει μια πολύ περιορισμένη εμβέλεια 100 μίλια γύρω από τη Μόσχα. Είναι όμως ένα σύστημα το οποίο έχει χρηματοδοτήσει η Ρωσία και όπου έχουν ξεκινήσει και όπου έχουν επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν ούτε οι Ρώσοι ξεκινάνε στον τομέα της αντιπυραυλικής άμυνας από το μηδέν έχουν ένα σύστημα το οποίο μπορεί να καταρρύψει ε, εξελιγμένα ε, βομβαρδιστικά, αλλά επίσης και ε, βαλιστικά βλήματα. Είναι κάτι σαν το Patriot 3. Θα φέρει λοιπόν αυτά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ρωσία, θα φέρει ε, και τα δικά της συστήματα η συμμαχία και το καλοκαίρι θα συμφωνήσουμε απόλυτα ποια θα είναι η σχέση μεταξύ του ρωσικού συστήματος και του συστήματος το οποίο έχει ως σκοπό να αναπτύξει ε, το ΝΑΤΟ. Ακολουθώντας βεβαίως τη συνηθισμένη προσέγγιση του ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ στην αντιαεροπορική άμυνα, δηλαδή πάντα υπό ε, την ανώτατη διοίκηση ε, του ΝΑΤΟ Ευρώπη και βέβαια λαμβάνοντας υπόψη ε, τα όσα θα πούν τα αρχηγεία που είναι αρμόδια για την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική άμυνα της Ευρώπης. Αυτά σας τα λέω για να σας εξηγήσω ποιες είναι οι ποια είναι τα αποτελέσματα της Λισαβόνας και ποιος πιστεύουμε πως είναι ο μελλοντικό μας ορίζοντας και επειδή ακούστηκε μια δήλωση την περασμένη εβδομάδα από τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων του δικού μας Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να το επαναλάβω γιατί είπε το Σεπτέμβριο του 2009 όταν ο πρόεδρος Ομπάμα αποφάσισε να αλλάξει ε, τα προηγούμενα σχέδια του Προέδρου Μπούς για ανάπτυξη αντιπυραυλικής άμυνας στην Πολωνία, πολλοί είπαν πως αυτό αλλάζει τη σχέση μας με τη Ρωσία. Άλλοι επέκριναν την απόφαση αυτή λέγοντας πως θα εκτροχιάσει τη σχέση μας με τη Ρωσία. Όμως, ο αντιπρόεδρος Biden μας είπε πως οι σκεπτικιστές αποδείχθηκε πως έκαναν λάθος. Στην Λισαβόνα συμφωνήσαμε ένα σχέδιο αντιπυραυλικής άμυνας ευρωπαϊκής με το ΝΑΤΟ και είδαμε πως υπάρχει βούληση για μια γρήγορη επικύρωση της συμφωνίας ΣΤΑΡΤ, όπως επίσης και για ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρώπη. Αποδείξαμε λοιπόν πως ο έλεγχος των εξοπλισμών και η αντιπυραυλική άμυνα μπορούν να συνδυαστούν. Merci, Bell. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέλ. Ο κύριος Λίζεκ, αντιπρόεδρος μας, θα ήθελε να μιλήσει από αυτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες και γι' αυτό θα μιλήσω στη γλώσσα μου, τα πολωνικά. Είμαι πολωνός, ε, δεν θα αναφερθώ όμως στα τελευταία επιχειρήματα που παρουσίασε ο κ. Πρέσβης. Ούτε θα αναφερθώ στον άλλο που έγινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από κάποιες οργανώσεις που γνωρίζουμε πολύ καλά τις τελευταίες μέρες. Θα ήθελα να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας του τομέα των πυράβλων. Αλλά βλέπει κανένας μια τεράστια διαφορά μεταξύ των σχεδίων που συζητήθηκαν και ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης της προηγούμενης κυβέρνησης, κυβέρνησης Μπούς δηλαδή, και αυτών που έχουμε εδώ σήμερα. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι η διαφορά κόστους του συστήματος που συζητάμε σήμερα. Αναφερθήκατε σε 200 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Προηγουμένως όμως, αν δεν κάνω λάθος, μιλάγαμε για δεκάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και θέλω να σε ρωτήσω, από πού προέρχεται αυτή η διαφορά. Δεν λέω ότι το πιο φθηνό προϊόν δεν δείχνει να είναι επίσης σοβαρό, αλλά εγώ από ό,τι κατάλαβα το θέμα είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν τα ισχύοντα συστήματα σε διάφορα κράτη-μέλη ΝΑΤΟ. Κατόπιν, μια που βρισκόμαστε εδώ σε ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω να αναφερθώ στο πώς βλέπει η Αμερική τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. και εκείνες τις χώρες που δεν είναι επίσημα μέλη του ΝΑΤΟ. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια είναι μέλη του ΝΑΤΟ, υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες που δεν ανήκουν. Πώς βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα της προστασίας και εκείνων των επικρατιών των χωρών που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Merci, Monsieur Σα ευχαριστώ. Να απαντήσετε. Ναι. Ε, δύο πάρα πολύ σημαντικέ και ενδιαφέρουσε ε, ερωτήσεις. Κόστος καταρχήν. Πριν από τρία χρόνια στα ΜΜΕ αναφέρθηκε ένα στοιχείο κόστους ότι η βαλιστική άμυνα της Ευρώπης ήταν 20 ε, δισεκατομμύρια ε, δολάρια. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η σχέση ισοτιμίας τότε, αλλά ήταν και περισσότερα από σήμερα. Τώρα βέβαια η διαφορά είναι τεράστια πραγματικά. Αλλά είναι σαν να προσπαθείτε να συγκρίνετε πορτοκάλια με ε, μήλα. <clears throat> Γιατί τα 20 της που είχαν αναφερθεί τότε προϋπόθεταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπάρχουν συνέβαλαν με τους ε, εξοπλισμούς που έχουν ήδη και ότι η Ευρώπη επίσης θα ξεκινούσε επίσης από το μηδέν. Επίσης προϋπόθεταν ότι η απέτηση ήταν για την άμυνα της επικράτειας του ΝΑΤΟ ε, κατά όλων των επιθέσεων από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Συμπεριλαμβάνει και της Βορειού παραδείγματος χάρη. Ή η δυνατότητα να υπερασπιστεί Γρυλανδία από μια επίθεση από την ε, Βόρειο Κορέα. Η, η πρόκληση λοιπόν, στην οποία βασίζεται αυτή η εκτίμηση, ήταν πάρα πολύ υψηλή. Επίσης, το θέμα της ε, κυβέρνησης Bush με την τρίτη ε, κατάσταση στην Παρουσία ήταν να συμβάλλει εθελοντικά η Αμερική για αυτή την τοποθεσία, την τρίτη αυτή τοποθεσία και το κόστος θα ήταν πολύ χαμηλότερο από τα 20 δις. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο χαμηλό όσο τα 200 εκατομμύρια για 10 χρόνια, αλλά θα ήταν πολύ πολύ χαμηλότερο. Η διαφορά ήταν όμως ότι το σχέδιο Bush ήταν να εγκατασταθούν αποκρουστές στην Πολωνία που θα μπορούσαν εκ μιας αρχής να αντιταχθούν σε ε, διπρωτικούς πυράβλους. Δηλαδή το ίδιο σύστημα ACBM όπως εκείνο που έβαλαν οι ΙΠΑ στην Αλάσκα και στην Καλιφόρνια. Με μια διαφορά φέροντας το τρίτο στάδιο. Κατά τα άλλα, πλήρως ικανό ε, άμυνα τύπου ACBM. Τώρα όμως, ε, ο στόχος αυτών των, ε, αυτών των εγκαταστάσεων ήταν να, προασ... να αμυνθούν στην Αμερική έναντι πυράβλων από τη Μέση Ανατολή. Τώρα όμως όλα αυτά τοποθετούνται στο πλαίσιο ΝΑΤΟ αν είχε προχωρήσει εκείνο το σχέδιο και δεν μπορούμε παρά να έχουμε κάνουμε εικασίε, το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να δει πώς θα συμπλήρωνε στην τρίτη πλευρά αυτό το σύστημα διπερωτικών ε, επιθέσεων με ένα σύστημα που θα κάλυπτε την Ευρώπη και από επιθέσεις από μικρότερες ε, τώρα έχουμε την κυβέρνηση Ομπάμα η οποία προτείνει συστήματα για μια άμυνα για το μεσοβελνικές και συμπλήρωση εάν και όποτε υπάρχει μια απειλή πραγματική για κάτι άλλο να συμπληρωθούν. Αυτή είναι δηλαδή μια σημαντική διαφορά όσον αφορά την βασική ιδέα, το βασικό σκεπτικό. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά κόστο. Η δεύτερη σα ερώτηση είναι πάρα πάρα πολύ ουσιαστική και πάει στην καρδιά του προβλήματος τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προσέγγιση της, την άμυνα και μάλιστα τη συλλογική άμυνα. Η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται να σα υπενθυμίσω εδώ εσά, προβλέπει σημαντικέ ρήτρε για τα θέματα αυτά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο της Συνθήκης Λισαβόνας είναι εκείνο που λέει ότι στην περίπτωση επίθεσης κατά της Ευρώπης, όχι δηλαδή η δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κονγκό ή δεν ξέρω πού αλλού, Παραδείγματο χάρη ε, αντιμετώπιση πειρατεία όπου τόσο καλά εργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, αλλά στην περίπτωση που υπήρχε μια επίθεση κατά τη Ευρώπη, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι επίση μέλη του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να στραφούν προ το ΝΑΤΟ για να του προσφέρει την οργάνωση της άμυνας. Θυμόσαστε ότι εγώ στην αρχή της παρέμβασης μου έθεσα την ε, απόφαση που ελήφθη στη Λισαβόνα για τους βαλιστικούς πυράβλους μέσα στο γενικό πλαίσιο της άμυνας, θα έλεγα ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, 21 είναι οι χώρες αυτές, θα ε, βασιστούν την ε, δομή του ΝΑΤΟ στην περίπτωση που υπάρχει πραγματικά μια τέτοια επίθεση κατά της Ευρώπης. Υπάρχει βέβαια μια πρόκληση τώρα για τις έξι εκείνες χώρες μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαντάζομαι ότι όσο αναπτύσσουμε το σύστημα θα έχουμε, όπως περιμένετε, διαβουλεύσεις με χώρες όπως την Σουηδία και τη Φιλανδία για να είμαστε σίγουροι ότι κατανοούμε πώς βλέπουν εκείνες τις εξελίξεις και τις δικές τους σχέσεις με το ΝΑΤΟ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ο κ. Ναυρονικόλας έχει το λόγο. Αντιπρόεδρος. We just a couple of points. I... Λίγες παρατηρήσεις, πρόεδρε. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στο τόσο χαμηλό κόστος. Και θέλω να ρωτήσω, ή εξακολουθεί να είναι ασφαλές το σύστημα αυτό με τόσο χαμηλό κόστος. Και ελέγχτε το σύστημα είναι ευέλικτο. Πεςτε μου υπάρχει μία ευρωπαϊκή συνιστόσα στο σύστημα αυτό. Θα είναι εύκολο δηλαδή για την Ευρώπη να ενταχθεί σε αυτό το μηχανισμό. Το επόμενο που θα θέλω να ρωτήσω. Όλοι ανησυχούν για την πυρηνική διάδοση. Ιδίω σε περιοχές του κόσμου δεν είναι πάρα πολύ σταθερές. Η ερώτησή μου είναι στις συνομιλίες με τη Ρωσία υπάρχει κάποια συνεννόηση για το θέμα αυτό. Οι συνομιλίες με την ε, Ρωσία βοηθούν να σταματήσει η διάδοση των πυρηνικών όπλων σε επικίνδυνες περιοχές του κόσμου ή τουλάχιστον σε χώρες που φαίνεται ότι θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνες αν αναπτύξουν ε, πυρηνικά όπλα. Τέλος. το μέλλον του αμυντικού συστήματος της Ευρώπης πώς το διαβλέπετε. Μας αναφερθήκατε σε τέσσερα στάδια μετά από χι χρόνια, αλλά αυτό το αμυντικό σύστημα θα είναι επαρκώς ικανό να αντιδράσει σε περίπτωση πυρηνικών επιθέσεων. Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ. Ο κύριος Λαντσπέργης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Είπα, Η είπα, αναρωτήθηκε ποτέ ή όχι, ποιοι είναι οι λόγοι η Ρωσία να επιθυμεί να διατηρήσει την Ευρώπη αδύναμη και όχι τόσο καλή στην άμυνά της ή να παραλύει τις δυνατότητες της άμυνας. Πώς βλέπετε τις ε, δράσεις της Ρωσίας και στην Ευρώπη, από τον Κάφκασο μέχρι την θάλασσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάγκελ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπέλ, μας ενημερώσατε για το νέο σύστημα με τον πιο ευνόητο τρόπο που έχω μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει το σύστημα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι που δεν αφαιρθήκατε μόνο σε στρατηγικές ανάγκες και επιχειρήματα, αλλά μας παρουσιάσετε και κάποιες πολιτικές σκέψεις. Πρόσφατα υπέβαλα εδώ στο σώμα μία ερώτηση προς ένα πολύ ψηλά ιστάμενο στρατηγό του ΝΑΤΟ αναρωτιόμενος κατά πόσον αυτό το σύστημα θα αυξήσει την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, ιδίως του Ισραήλ. Γιατί εσείς δεν αφαιρθήκατε αυτή τη χώρα που μας ανησυχεί περισσότερο και για την οποία χρειαζόμαστε αμυντικά συστήματα. είναι νομίζω προφανές για όλους που είναι εδώ στην αίθουσα ποια είναι η λόγω χώρα που μας ενδιαφέρει. Η χώρα αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας όσον αφορά ιδίως την ε, σύγκρουση Παλαιστινίων Ισραηλινών. Εγώ πιστεύω στη διπλωματία. Παρά αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Που βέβαια παρουσιάζει τις αδυναμίες γενικά της ε, διπλωματίας. Παρ' όλα αυτά για μένα αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση. Διπλωματική εργασία, διπλωματική αναζήτηση λύσεων για οποιοδήποτε πρόβλημα. θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο θα πρέπει να αυξήσει την ασφάλεια του Ισραήλ. Και αν αυτό αληθεύει, θα αυξήσει και την πρόθεση, την βούληση του Ισραήλ να επιληθούν τα προβλήματα με τους Παλαιστινίους ειρηνικά και επικοδομητικά. Και θα πρέπει επίση να αλλάξει την γενική ατμόσφαιρα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς προωθώντας την βούληση συμβιβασμών και την ελληνική προσέγγιση. Σφάλω. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριος Κυρίλοφ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω πως άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα είπατε. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα. Να μου πείτε αν είναι τεχνικά βιώσιμη αυτή η συνεργασία με τη Ρωσία. Εσείς αναφερθήκατε σε κάποιες ε, προσπάθειες που έχουν γίνει με προσωμιώσεις, με ασκήσεις μέσω υπολογιστή και μιλήσατε για μια ενδεχόμενη ρωσική συνεισφορά. Έχουμε το σύστημα αντιπεριβλακής άμυνας της Μόσχας κτλ. Όμως το θέμα αυτό είναι πολιτικά εξαιρετικά καυτό, ευαίσθητο, αλλά παράλληλα, ενώ πολιτικά έχει βρεθεί μια λύση, είναι και τεχνικά εξαιρετικά δύσκολο. Μέχρι τον Ιούνιο λοιπόν του 2011 θα έχετε καταφέρει να λύσετε τις τεχνικές παραμέτρους αυτής της συνεργασίας. Εδώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος πως αυτό μπορεί να συμφωνηθεί ε, και θα ακούσουμε και τον κύριο Ρογκόζιν αργότερα. Πείτε μου λοιπόν πώς λοιπόν τα υπολείμματα ε, τις ανταγωνιστικές σχέσεις που είχαμε και αυτή της έλλειψης εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τα δύο μέρη θα ε, τα υπερβούμε έτσι ώστε να περάσουμε σε πια μία πιο εξελιγμένη μορφή αυτού του συστήματος γιατί ενδεχομένως τα δύο μέρη θα θελήσουν να κρατήσουν κάποια από τα τεχνικά τους επιτεύγματα κρυφά. Γι' αυτό σας ρωτώ πολιτικά πώς θα τα καταφέρουμε. Γιατί αν βεβαίως αυτή η δοκιμή που θα κάνουμε αποτύχει, ίσως τελικά αυτό ε, να μας οδηγήσει σε μια οπισθοχώρηση σε σχέση με το όσο έχουμε επιτύχει στο μέλλον. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κύριο Μπέλ για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί άκουσα πολλές ερωτήσεις. Να σας πω πως για το θέμα της ασφάλειας πρέπει να υπογνωρίσουμε πως αυτή αυτή, αυτά τα αναχαιτιστικά βλήματα έχουν ως σκοπό να πλήξουν εισερχόμενους πυράβλους ε, που δεν φέρουν είτε συμβατικές είτε πυρηνικές κεφαλές γιατί αν εκτοξευθεί κατά λάθο αυτός ο πύραυλος, που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, νομίζω ότι απλώς θα εκτοξευθεί στην ατμόσφαιρα και εκεί θα καεί. Μιλάτε λοιπόν για τα ανεχετιστικά AIDS που έχουμε πάνω στους κρούς, πυράβλους κρούς και αυτό έχει αποδειχθεί από τα πειράματα που έχει κάνει το Αμερικανικό Ναυτικό χωρίς να έχουν υπάρξει ατυχήματα που θα οδηγήσουν σε ανησυχίες περί ασφάλειας, πώς τα καταφέρουν θαυμάσια. Και αυτό ισχύει ε, και για την αντιπυραυλική άμυνα περιοχής ε, που, έχουν, ε, που έχει εγκατασταθεί στην Πολωνία και στη Ρουμανία ή που θα εγκατασταθούν εκεί. Εκεί πρέπει να σας πω πως αυτά τα αναχαιτιστικά δεν φέρουν ε, εκρηκτικά με αποτέλεσμα ε, να μην ε, δημιουργούν πρόβλημα. Για τους αναχαιτιστικούς πυράβλους μικρής εμβέλειας πρέπει να σας πω πως χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια χωρίς πρόβλημα. Ε, πέραν του συστήματος ε, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από κοινού για το LTBMD, να σας πω πως το μενού το οποίο προσφέρεται σε επίπεδο στρατιωτικών δυνατοτήτων είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Τα κράτη της συμμαχίας μπορούν να επιλέξουν, εάν το επιλέξουν, να συνεισφέρουν την εθνική τους ε, συνεισφορά στο συνολικό αρχιτεκτόνιμα του ΝΑΤΟ. Και στο πρόγραμμα ALTBMD, δηλαδή Επιχειρησιακής Αντιπυραυλικής Άμυνας, ε, τέλη της χρονιάς θα δείτε πως θα αναπτύξουμε μια μεγάλη γκάμα συμμαχικών δυνατοτήτων που έχουν ε, υποστηριχθεί από την ευρωπαϊκή τεχνολογία, το τάλις κτλ. Θα σας τα παρουσιάσω νομίζω αργότερα έχετε το σύστημα Astor που είναι Ιταλογαλλικό, έχετε το Ολλανδογερμανικό των Patriot, έχετε τις ε, φρεγάτες ε, ε Ισπανικές που μπορούν να φέρουν τέτοιου είδους πυράβλους και έχετε και Γαλλογερμανική Ιταλική συμμαχία, το NIAD, e ε, που προσφέρει δυνατότητες ε, αεροπορικής αντιπυραυλικής άμυνας. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι δυνατότητες ε, μικρότερης εμβέλειας TMD που αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί και στην Ευρώπη και που έχουν αποδεδειγμένα φανεί πως είναι διαλειτουργικές με το, με το κέντρο διοίκησης ε, και χειρισμού του ALTBMD του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν μπορούν να τοποθετηθούν στη νέα στρατηγική που καθορίζει το ΝΑΤΟ για την αντιπυραυλική άμυνα. Αν λοιπόν οποιοδήποτε από τους συμμάχους ή από τα Υπουργεία Άμυνας της Συμμαχίας αποφασίσουν να χρηματοδοτήσουν τα upper layer ε, όπλα, ξέρω από την προσωπική μου εμπειρία πως οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν σχέδια στα σκαριά, έχουν κάνει κάποια έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο αυτό και το μόνο που χρειάζονται είναι χρηματοδότηση για την παραγωγή. Βέβαια, καταλαβαίνετε, λόγω τη χρηματοπιστωτική κρίση αυτό μάλλον δεν είναι πιθανό. Αλλά εάν οποιοδήποτε από τους συμμάχου μου στο ΝΑΤΟ, μου στο ΝΑΤΟ θέλουν να επενδύσουν εθνικά στα δικά τους προγράμματα, έτσι ε, να χρησιμοποιήσουν ε, την χαμηλότερη γκάμα δυνατότητα TMD που έχει ήδη αναπτυχθεί και να προσπαθήσουν να καλύψουν μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή ε, με αντιπυραυλική άμυνα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε πολιτικό, ούτε τεχνολογικό, ούτε στρατιωτικό. Γιατί μπορούν, επαναλαμβάνω, τα συστήματα αυτά να ενταχθούν στο σύστημα του ΝΑΤΟ ε, στα πλαίσια, ε, με τον ίδιο τρόπο μάλλον που θα ενταχθεί η phased adaptive προσέγγιση, δηλαδή αυτή η σταδιακή προσαρμογή για την Ευρώπη. Τώρα, για τη σχέση με τη Ρωσία και το θέμα της διασποράς, Νομίζω πως θα πρέπει ο κύριος Πρέζης να μας απαντήσει γιατί είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον για τη Ρωσία αλλά νομίζω πως το ρεκόρ της Ρωσίας είναι εξαιρετικά θετικό ε, και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν απευθύνει πολύ συχνά ευχαριστήσεις προς τη Ρωσία η οποία τα τελευταία χρόνια υπερψηφίζει τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών με στόχο να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει ε, πυρανικά όπλα και νομίζω πως ήταν σημαντική η βοήθειά της και είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου που το Ιράν αντιμετώπισε αυτό το στεναρό μέτωπο σε επίπεδο ε, Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. οι Ηνωμένε Πολιτείε και κυρίω με αυτή την ε, επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία που προωθεί ο πρόεδρο Ομπάμα, προωθούν ε, το θέμα αυτό τη μη διασπορά. Ακούστηκε και μία ερώτηση για να μείνουμε στις σχέσεις με τις ε, Ρωσία. Νομίζω πως το θέμα ήταν για ποιο λόγο θέλει η Ρωσία να διατηρήσει το ΝΑΤΟ αδύναμο και σε παράλυση στο θέμα της αντιπυραυλικής άμυνας. Πρέπει να σας πω πως με συγχωρείτε, διορθώνω, θέλει να κρατήσει αδύναμη και σε παραλυσία την Ευρώπη. Νομίζω πως εμείς ε, κάναμε ένα βήμα μπροστά στη Λισαβόνα, γιατί έχουμε ένα νέο δικό χάρτη για τη συνεργασία στην αντιπυραυλική άμυνα με τη Ρωσία και νομίζω πως οι συζητήσεις που θα γίνουν με σοβαρότητα τις επόμενες εβδομάδες ε, είναι ενδιαφέρουσες. Έχω πολλές προσδοκίες και αναμένω μια συμφωνία η οποία ελπίζω θα έχει ε, σχεδιαστεί στη μέχρι τον Ιούνιο. Βέβαια το πρόβλημα είναι πάντα οι λεπτομέρειες και δεν θέλω να υποβαθμίσω τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε με κάποια από τα θέματα αυτά. η οι Ρώσοι ομολογοί μας έχουν τονίσει ε, το πρόβλημα του επιμερισμού του κόστους ε, και της τεχνολογίας ε, σε περίπτωση που έχουμε μεταφορά ή όχι τεχνολογίας. Είναι θέματα σημαντικά. Όμως, εγώ αισθάνομαι αισιόδοξο γιατί ω αξιωματούχο του ΝΑΤΟ ε, αυτή την, την περασμένη δεκαετία συνεργάστηκα πολύ επιτυχώ με τη Ρωσία και το είπα και προηγουμένω. Μετά άκουσα και μία ερώτηση για τη σχέση μεταξύ της αντιπυραυλικής άμυνας και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και βεβαίως εδώ ακούστηκε και το θέμα της διαπραγμάτευσης Παλαιστινίων Ισραηλινών, όπως επίσης και το θέμα του Ιράν. Η άποψή μου είναι πως εδώ και χρόνια η αντιπυραυλική άμυνα είναι μια, ένα βοήθημα, αλλά δεν αποτελεί τη λύση. Γιατί η λύση θα προέρθει μόνο από την στεναρή διπλωματία. Όμως η αντιπυραυλική άμυνα βοηθάει με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα τα έθνη τα οποία έχουν αντιπυραυλική άμυνα αισθάνονται πιο ασφαλή. δεν αποτελούν ε, υποκατάστατο, αλλά με την αντιπυροβλική άμυνα έχετε περισσότερες δυνατότητες για να αντιμετωπίσετε μια κρίση. Για μένα λοιπόν ήταν σημαντικό το ότι η διοίκηση Bush το επιβεβαίωσε πριν από τρία χρόνια σε κάποιες από τις περιοδικές κρίσεις που αντιμετωπίσαμε με τη, με τη Βόρειο Κορέα για τις πυρηνικές της προσπάθειες, πως επειδή το αντιπυραυλικό σύστημα στην Αλάσκα και στην ε, Καλιφόρνια ήταν πλέον λειτουργικό, είχαν περισσότερο χρόνο για να επιδιώξουν διπλωματικές λύσεις για την κρίση αυτή. Δική μου λοιπόν άποψη είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αντιπυραυλική άμυνα για να αγοράσουμε χρόνο έτσι ώστε να κάνει κάποιες προσπάθειες η διπλωματία. Υπάρχει, δεν θα πω παραπάνω, μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ των επιλογών που κάνει κανείς κάποια στιγμή κρίσης, αλλά πιστεύω πως σε κάποιο βαθμό η η επιχειρησιακή αντιπυραυλική άμυνα, και αυτό μπορείτε να το δείτε και αλλού, μπορεί να βοηθήσει. Ελπίζω επίσης πως αυτή η αντιπυραυλική άμυνα και η απόφαση του ΝΑΤΟ να συνεχίσει τις προσπάθειες εδώ, σε συνεργασία πάντα με τη Ρωσία, δεδομένης της δεδηλωμένη ανησυχίας της Ρωσίας για την διασπορά αυτών των πυράβλων και τις ανησυχίες που έχει εκφράσει για τα προγράμματα ανάπτυξης ε, πυράβλο του Ιράν μας οδηγεί στο να στείλουμε ένα μήνυμα μέσα των αποφάσεων αυτών στο Ιράν πως οποιαδήποτε προσπάθεια που θα κάνει ε, για να βρει ε, δυνατότητα παράδοσης πυρηνικού όπλου ε, κάποιας εμβέλειας δεν θα λειτουργήσει σε μελλοντική κρίση. Για το λόγο αυτό λοιπόν έχω να σας πω πως για την πυραυλική άμυνα μπορεί να βοηθήσει ως αποτροπή. Δεν θέλω βέβαια να συνεχίσω σε αυτή τη λογική, αλλά πιστεύω πως θα δώσει μια διπλωματική δυνατότητα να λυθούν τα προβλήματα αυτά με κάποιο άλλο τρόπο. Uh, θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι υπάρχει μια, τεχνικά αυτή μέθοδος για τη συνεργασία και θα ήθελα να αναφερθώ στην εμπειρία που είχα 2002-2008 με το πρόγραμμα TMD για τη σχέση με τη Ρωσία, γιατί οι ιδέε που είχαν υιοθετηθεί τότε δεν είχαν σαν στόχο να υπάρχει ένα ενιαίο συνδυασμένο σύστημα ε, άμυνας πυράβλων. Υπήρχε μια ευρεία βάση διαλειτουργικότητας ένωσης δηλαδή των δυναμικών και ταυτόχρονα όσον αφορά το TMD ΝΑΤΟ-Ρωσία, η ιδέα που ακολουθήσαμε ήταν ότι έχουμε ανεξάρτητα μεν, αλλά συντονισμένα συστήματα άμυνας. Και το ένα δίπλα στο άλλο και το κάθε πλευρό θα ήταν υπεύθυνο, η κάθε πλευρά θα ήταν υπεύθυνη για την λήψη αποφάσεων στον τομέα που είχε σαν στόχο να προστατεύσει. Στην τελευταία ε, γυμνάσια που έγινε το Γενάριο του 2008, ήρθαν οι Ρώσοι στο ΝΑΤΟ πριν από μερικέ εβδομάδε και είχαν μια πολύ καλή παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το ΝΑΤΟ και η Ρωσία σε ένα υποθετικό σενάριο για την πολιτεία του Άινταχου και άμυνα κατά πυράβλων προχώρησαν από το βορρά. Και εκεί κάθε πλευρά είχε τη δική της ανεξαρτησία, αυτονομία, αλλά επειδή οι ζώνες άμυνας ήταν η μια δίπλα στην άλλη, η συνολικά προστατευόμενη περιφέρεια ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και μάλιστα μια φορά ε, που κάνανε μια άσκηση κατά την οποία ε, έγινε επίθεση σε ένα κέντρο πολύ πολύτιμο στην περιφέρεια που προστάτευε το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ δεν είχε πια αμυντικούς πυράβλους και επικοινώνησε με τη Ρωσία και είπε μπορείτε εσείς να καλύψετε αυτή, αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και είπανε ναι. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα συνεργασίας ακόμα και αν δεν υπάρχει ανταλλαγή τεχνολογικών συστημάτων, ολοκλήρωση των συστημάτων, εναρμόνιση των συστημάτων μέσα στα πλαίσια των δύο πλευρών. Εμείς θα συνεχίσουμε την ε, συνεργασία TMD σαν πρώτο βήμα κάτω από την ε, Συμφωνία του Λισαβόνας και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να Αναφερθούμε ακριβώ σε αυτή την τόσο επιτυχή ε, δοκιμή του Ιανουαρίου του 2008 για να δούμε πώ γίνεται η συνεργασία των ΜΕΝ και των ΔΕ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε κάθε ερώτηση και τώρα θα συνεχίσουμε με τη δεύτερη ομάδα ομιλητών. Ο κύριος Ρογκοζίν, ε, πρέσβης στο ΝΑΤΟ της Ρωσίας, έχει το λόγο. Bien, Monsieur l'ambassadeur, bienvenue euh, à cette sous-commission. Euh, Καλώς ορίσατε. Ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ, γιατί όπως είπε και ο κύριος Μπέλ προηγουμένως, φαίνεται πως ε, στη σύνοδο ή στις συνόδους καλύτερα της Λισαβόνας καταφέραμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σε σχέση και στις σχέσεις μας με την Ρωσία. Θυμόσαστε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μία από τις γνωμοδοτήσεις του πέρσι ε, εκφράστηκε υπέρ μιας, ε, ενός διυπηρωτικού διαλόγου, έτσι το είχαμε χαρακτηρίσει. Και ξέρετε ότι υπήρχαν δυνατότητες ε, αναρώτησης πώς θα ήταν δυνατή μια συνεργασία, ένας διάλογος με τη Ρωσία χωρίς να περάσουν κάποια πρώτα στάδια πάρα πολύ σημαντικά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας να ακούσουμε τη δική σας άποψη, την άποψη της Ρωσίας δηλαδή, για τι εξελίξει αυτές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην ε, σημερινή ακρόαση για να πάρω το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω πως θα καταφέρω και να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας παρακαλώ να μου συστήνεστε ε, έχω συνηθίσει να συνεργάζομαι με τους, με τους βουλευτές στην Τούμα στη Ρωσία. Ήμουν ο ίδιος ε, βουλευτής, ήμουν αντιπρόεδρος της ε, Τούμα στη Ρωσία και πρέπει να σας πω πως πάντα με ιδιαίτερο σεβασμό αντιμετωπίζω την κοινοβουλευτική διπλωματία. Ξέρω πως στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να σταθώ ως άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τη σημασία του διαλόγου με την ε, κοινωνία και κατανοώ πόσο σημαντική είναι η κοινωνική στήριξη προσπάθειας που κάνουμε και τα αντιμετωπίζω αυτά όχι σαν επαγγελματίας διπλωμάτης. Θα ήθελα να σας πω πως το σύστημα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που είναι η αντιπυραυλική άμυνα, ε, πρέπει να σας πω πως ασχολήθηκα με αυτό στο διδακτορικό μου, που είχε να κάνει με ε, το θέμα της ε, γαλλικής άμυνας και ε, αυτό ήταν και το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη, ευχαριστημένος που άκουσα τον κύριο Μπέλ, ο οποίος με πολύ σοβαρότητα και σε ιδιαίτερο βάθος εξήγησε ακριβώς τι συμβαίνει στο θέμα αυτό και παρουσίασε την άποψη του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα επίσης να πω πως εγώ στεναρά στηρίζω τη συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας και νομίζω ότι σε όλους τους χώρους που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε έχουμε αποθέματα και κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τη συνεργασία μεταξύ Δύσης και Ρωσίας στα θέματα της άμυνας και όχι μόνο στα θέματα άμυνας. Ε, έχουμε ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα ε, πρέπει να σας πω που περάσαμε και μία φάση αρκετά δύσκολη, γιατί αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μας είναι πολύ πιο ε, είναι ιδιαίτερα ε, σφιχτές και πρέπει να σου πω πως είναι πλέον δύσκολο να θέσει κανείς υπό αμφισβήτηση αυτή τη συνεργασία. Το θέμα λοιπόν αυτό της αναχέτησης των πυράβλων μικρής εμβέλειας είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια πραγματικά βαθιά συνεργασία με τις χω... μεταξύ των χωρών μας και μετά τα όσα ακούσαμε και στην Σύνοδο της Λισαβόνας αλλά και στη Σύνοδο ΝΑΤΟ-Ρωσίας θα πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Θα ήθελα να εξετάσουμε στα πλαίσια αυτού του προβλήματος μια διαφορετική άποψη, έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι αμφιβολίες και αμφισβητήσεις που ακούγονται και στην Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αν θυμόσαστε, το δόγμα αυτό της αντιπυραυλικής άμυνας ε, εκφράστηκε για πρώτη φορά από τον πρόεδρο Μπούς τον νεότερο, όπου η κατάσταση ήταν η εξής. Αυτή τη στιγμή θα είχαν αποφασίσει, τότε είχαν ε, είχαν ε, ε, επιλέξει τρεις ε, τόπους εγκατάστασης στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη. Η Πολωνία έχει ζητήσει την εγκατάσταση 10 τέτοιων αναχαιτιστικών ε, εγκαταστάσεων. Η Τσεχία είχε ζητήσει να εγκατασταθούν τα στρατηγικά ραντάρ εξ διαπασών, τα οποία κατά τη γνώμη των ε, Ρώσων εμπειρογνωμών θα μπορούσαν να ε, φτάσουν οι εκτοξεύσεις από εκεί και την ρωσική επικράτεια, αλλά θα μπορούσε, ο σκοπός τους βασικός ήταν η εξασφάλιση από την ρωσική επίθεση. Βεβαίως, είχε χρησιμοποιηθεί τότε ως πρόφαση η απειλή που παρουσιάζει το Ιράν αλλά τότε εμείς είχαμε εκφράσει ανησυχίες για το κατά πόσο στοχοποιείται το Ιράν με τον τρόπο αυτό και θεωρούσαμε πως έγινε μια προσπάθεια εξουδετέρωσης ε, του, ε, της, ε, του στρατη, της στρατηγικής άμυνας της ίδιας της Ρωσίας. Μετά ε, που άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, άλλαξε και η κατάσταση και η νέα διοίκηση των ΗΠΑ, με την οποία συνεργαζόμαστε πολύ στενά και όπου πιστεύουμε πως ο πρόεδρος Ομπάμα ε, για τις ε, ρωσοαμερικανικές σχέσεις είναι μια μεγάλη ευκαιρία γιατί είναι ένας άνθρωπος ρεαλιστής, ο οποίος έχει σκοπό να λύσει προβλήματα όχι μόνο άμυνας, αλλά και θέματα πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας. Πιστεύουμε λοιπόν πως αυτή η νέα αμερικανική ε, διοίκηση ανασκεύασε τα διάφορα προγράμματα επιχειρησιακής αντιπυραυλικής άμυνας Ε, και θα ήθελα να εκφραστώ για κάποιες φοβίες οι οποίες κατά καιρού έχουν ακουστεί για το θέμα αυτό. Καταρχήν, για το σύστημα αυτό της αντιπυραυλικής άμυνας. Όντως, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή πυραμίδα ε, δράσεων δυνατοτήτων είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος επιχειρησιακής πυραυλικής άμυνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σφαιρικά. Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για το ευρωπαϊκό σκέλος. Αυτό αποτελεί ένα μόνο βήμα για την οικοδόμηση και των υπολείπων. Εάν στο παρελθόν σύμφωνα με τα σχέδια του Μπούς μιλούσαμε για την εγκατάσταση ρεντάρ στη Τσεχία και την Πολωνία και είχαμε για το θέμα αυτό αρκετές αμφιβολίες, πρέπει να σας πω πως αντίθετα για το νέο σύστημα πιστεύουμε πως το σύστημα αυτό είναι απόλυτα κινητό, είναι φορητό, άρα δεν μπορεί, δεν μπορεί να προβληθεί το... Αυτά τα αναχαιτιστικά ή εκτοξευτήρες που θα βρίσκονται σε σκάφη που θα πλέουν στις νότιες θάλασσες, δεν δίνουν καμία εξασφάλιση πως τα πλοία αυτά δεν θα αλλάξουν τον τόπο στον οποίο πλέον και θα μπορούσαν πραγματικά να βρεθούν κάπου διαφορετικά και να στοχεύουν κάποιον άλλο. Αυτή λοιπόν η φορητή ε, επιχειρησιακή αντιπυραυλική άμυνα μου θυμίζει την όπερα Φίγκαρο. Φίγκαρο εδώ, ο Φίγκαρο εκεί. Και κανείς αυτή τη στιγμή δεν προτίθεται να περιορίσει το μέρος εγκατάστασης αυτών των πυράβλων. Αν λοιπόν μιλάμε για για, συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, τότε γιατί να μην περιορίσετε ε, την επιχειρησική αντιπαρευλική άμυνα σε κάποιους με κάποιε παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, γεωγραφικές συντεταγμένε, Να δίνετε συντεταγμένε, όπου θα λέτε ότι εκεί θα βρίσκονται αυτοί οι πύραυλοι αναχαιτιστικοί και μόνο. Δεύτερον, περιορισμό θα πρέπει να γίνεται και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στιμάτων που θα αναπτυχθούν. Εάν μιλάμε για την ανάγκη αναχέτησης πυράβλων μικρής και μέσης εμβέλειας, και νομίζω οι Αμερικανοί φίλοι μόνο σε αυτό αναφέρονται και οι πυρογνωμονές τους, τότε αυτή η αναρχιτιστική πύραυλη θα πρέπει να έχουν κατανεμηθεί ανάλογα με την απειλή. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν διυπηρετικού πυράβλους, γιατί δεν διαθέτει τέτοιους στο Ιράν. Ούτε κάποια άλλη χώρα που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνική τεχνολογία. Αυτή λοιπόν η διπυρωτική πύραυλη ανήκουν σε μια μικρή ομάδα ε, ε, κρατών, την πυρηνική πεντάδα και ξέρετε πως πολλές φορές τη ρωσική αρκούδα την ανησυχεί το ότι την πειράζουν και προσπαθούν ε, να την ενοχλήσουν εκεί που κοιμάται. Είναι λοιπόν στο δάσος και έρχονται 28 κυνηγοί που είναι τα 28 κράτη του ΝΑΤΟ και λένε «Αρκούδα, έλα να γίνουμε φίλοι και έλα να κυνηγήσει μαζί μας λαγούς». Και η Αρκούδα χαίρεται που την κάλεσαν να κυνηγήσει μαζί τους 28 κυνηγοί και τότε ξαφνικά να ρωτιέται και γιατί οι κυνηγοί αυτοί φέρουν ε, αυτή τη στιγμή όχι καραμπίνες για να κυνηγήσουν λαγούς, αλλά ε, οπλισμό που κάνει μόνο για αρκούδες. Τώρα για τα 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα χρειαστούν για να χρηματοδοτήσει το σύστημα, εγώ θα είμαι ειλικρινή μαζί σα. Πραγματικά αμφιβάλλω πω χρειάζονται μόνο 200 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ νομίζω πω με 200 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να γυρίσει κανεί ταινία στο Hollywood ε, για την αντιπυραυλική άμυνα, όχι κάτι παραπάνω. Για να στήσει κανεί πραγματική αντιπυραυλική άμυνα επιχειρησική, μιλάμε για δι επί δολαρίων. Βέβαια το θέμα εδώ είναι για την προσαρμοσμένη στρατηγική η οποία σε φάσεις θα εξαπλωθεί και θα αναπτυχθεί πάνω από την Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε για μια διασύνδεση τεχνολογίας η οποία ήδη υφίσταται στην επικράτεια των ευρωπαϊκών χωρών και που έχει ήδη αναπτυχθεί ή για ε, αμερικανική τεχνολογία την πυραυλική που έχει αναπτυχθεί από τους ε, Αμερικάνους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έτσι λοιπόν μιλάμε όχι για αμφιβολίες αλλά για θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Ξέρετε, πως οι Ευρωπαίοι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν τέτοιου είδους ε, επιχειρησιακή αντιπυραυλική άμυνα. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για νατοική επιχειρησιακή αντιπυραυλική άμυνα, μιλάμε για αμερικανική τεχνολογία η οποία θα αναπτυχθεί στην ευρωπαϊκή επικράτεια με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Διαχείριση, χειρισμός, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή αυτή της άμυνας θα γίνεται από το ΝΑΤΟ. Χειρισμός λοιπόν και διοίκηση. Από τον αρχηγό επιτελείου του ΝΑΤΟ, που αυτή τη στιγμή είναι και αρχηγός επιτελείου των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Άρα λοιπόν, να το πω πιο απλά. Βεβαίως, είναι ένα τοικό το σύστημα, αλλά το κουμπί θα το πατάνε οι Αμερικάνοι. Τι σημαίνει αυτό. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η πλασματική απειλή, η οποία θα μετατραπεί σε με πραγματική απειλή. Θα γίνει μία συνάντηση στο ΝΑΤΟ, θα γίνουν κάποια, ε, κάποιες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και εκείνη τη στιγμή οι Ευρωπαίοι θα θελήσουν να εξουδετερώσουν αυτή την απειλή και δεν θα χρειαστεί να εμπιστευτούν μόνο το ΝΑΤΟ, αλλά συγκεκριμένα τα αμερικανικά συστήματα αναχαιτιστικών πυράβλων που έχουν στα χέρια τους οι Αμερικανοί, όχι το ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνω. Ο κύριος Μπέλ είπε ότι μέχρι το 2020 η άμυνα αυτή θα έχει τη δυνατότητα ε, της αναχέτησης των διεπηρετικών πυράβλων. Και τότε ρωτώ το εξής. Γιατί εμείς σήμερα είμαστε σε ομοιρία και δαιμονοποιούμε το Ιράν. Γιατί συζητάμε για το θέμα της απόκτησης πυρηνικής τεχνολογίας από το Ιράν, πυραυλικής ε, τεχνολογίας και άλλων είδων στρατιωτικών τεχνολογικών. Ποιος είναι ο λόγος. Είναι όντως το Ιράν η χώρα η οποία έχει στόχο να επιτεθεί στην Ευρώπη. Πέρσι η οι εμπειρογνώμονε τη Ρωσία, τη Ευρώπη και τη Αμερική, στα πλαίσια του Συμβουλίου ε, ΝΑΤΟ-Ρωσία, μίλησαν για τι απειλέ ε, που, απειλούν, που μας απειλούν και αυτά τα είδαμε ήδη από το Δεκέμβριο πέρσι. Στην Λισαβόνα αποφασίστηκε και το θέμα αυτό της επιχειρησιακής αντιπυραυλικής άμυνας. Έγινε και μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών για να δοθούν κάποιες ε, ε, εκτιμήσεις και να γίνουν κάποιες αξιολογήσεις για την στρατηγική ασφάλεια με έγγραφα τα οποία είναι απόρριτα. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, να σας πω όμως πως τα θέματα τα οποία ε, αναφέρονται στο θέμα αυτό το πυραυλικό δεν καταφέραμε εδώ να ε, λιάνουμε όλα τα προβλήματα. Δεν μπορεί κανείς να τετραγωνίσει τον κύκλο και αποφασίσαμε να δεχτούμε το ότι διαφωνούμε και να παρουσιάσουμε ένα μνημόνιο με τα σημεία διαφωνίας. Μιλάμε για θέματα τα οποία έχουμε κρίνει αντικειμενικά, γιατί καθένας από εμά έχει βέβαια τις εμπειρογνώμονές τους με τις δικές του θέσεις, με τα δικά του εθνικά στοιχεία, με τα δικά του ε, ε, με, τα, με τις δικές του μυστικές προφορίες και δόξα θα οι δικές μας μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν ακόμα. Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θεωρεί πως είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βρούμε ποιος είναι ο κακός της υπόθεσης. Ούτε μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε την απειλή αυτή των πυραυλικών επιθέσεων. Βεβαίω πρέπει να συνεχίσουμε τι πολιτικέ προσπάθειε συνεργασία με την Τεχεράνη για να την πείσουμε πώ μπορούμε να τη προσφέρουμε κάποια εχέγγυα έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνει αυτή την κούρσα εξοπλισμό που βέβαια παρασύρει και κάποιους άλλους από τη διεθνή κοινότητα. Στη Λισαβόνα συμφωνήσαμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτή την εταιρική στρατηγική σχέση και όντως έχουμε τη βούληση. Τι σημαίνει πραγματική εταιρική σχέση. Όταν αντιμετωπίζουμε τους εταίρους μας με σεβασμό, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου διαφωνεί μαζί μας, ακόμα και όταν έχει φοβίες και ανησυχίες, επειδή ακριβώς είναι θέματα ασφάλειας και καταλαβαίνετε όλοι έχουμε την ιστορία μας, τα προβλήματα της χώρας μας, έχουμε διαφορετικές σχέσεις μεταξύ μας. Η εταιρική σχέση είναι αυτή κατά την οποία σέβεσαι όχι μόνο τα όσα εμπίπτουν στην κοινή αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων ασφάλειας, αλλά και των θεμάτων στους οποίους υπάρχει σε οποία υπάρχει διαφωνία. Δηλαδή πρέπει να σεβόμαστε και τους φόβους των εταίρων μας. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της Ευρωπαϊκής Επιχειρησιακής Αντιβρακής Άμυνας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα ήθελα εσείς να καταλάβετε ποιοι είναι οι περιορισμοί, πραγματικοί περιορισμοί για τη Ρωσία. Θα θέλαμε όντω να έχουμε κοινέ παραμέτρους ασφάλειας και κυρίως προς την κατεύθυνση ε, που θεωρούμε πως θα έχουμε απειλές, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα λένε οι πυρογνώμονές μας. Ε, εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω, ούτε χρειάζεται να παρακολύσουμε τους εταίρους μας από τα όσα επιθυμούν να κάνουν. Ε, ποιος απειλεί τη Βόρεια Ευρώπη, την Ευρώπη του Βορρά, ποιος την απειλεί. Η Ιρλανδία, η, η Σουηδία, ε, με συγχωρείτε, η Λευκή Αρκούδα, η Πολική Αρκούδα και εκεί αμφιβάλλω. Το σύστημα λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθεί στα σημεία για τα οποία υπάρχουν ενδεχόμενες απειλές. Εάν λοιπόν η Ρωσική Ομοσπονδία μέσω αυτής της συνεργασίας και ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με το, ΝΑΤΟ διαπιστώσει πως δίπλα στα βορειοδυτικά μας σύνορα ε, εμφανιστούν τέτοιου είδους πυραυλικά ε, συστήματα αναχέτησης που εξασφαλίζουν την ασφάλεια της Ευρώπης στο Νότο κατά τις δικές σας απόψεις, αλλά κατά τη γνώμη των δικών μας εμπειρογνωμόνων έχουν ως σκοπό να περιορίσουν την ε, ε, επιθετική δυνατότητα και δυναμικό που έχει η Ρωσία, τότε θα διαταράξει μια ισορροπία την οποία έχουμε χτίσει εδώ και χρόνια. Και δεν νομίζω πως από επιθυμούν κάτι τέτοιο οι Αμερικανοί συνάδελφοι. Γιατί για μας αυτό θα αποτελέσει σημείο ανησυχίας και θα είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστούμε με εσά εάν πιστεύουμε ότι η ασπίδα αυτή έχει στραφεί εναντίον μας. Εμεί δεν θεωρούμε πω το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι μοναδικό. Το ρωσικό σύστημα ανεχταστικών πυράβλων είναι υπό την εθνική κυριαρχία έλεγχο και διοίκηση. Βεβαίω σεβόμαστε το ΝΑΤΟ, είναι μια συμμαχία κυρίαρχη η οποία ελέγχει το δικό της και διοικεί το δικό της σύστημα ε, αντιπυραυλικής άμυνας. Και νομίζω θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν δύο υπότες στέκονται πλάτη-πλάτη και προσπαθούν ο καθένας να βοηθήσει τους δικούς του. Αν λοιπόν κάποιος πύραυλος περάσει μέσα από τη δικό μας ε, αεροπορικό χώρο και στοχεύει την ρωσική επικράτεια ή τις ευρωπαϊκές ε, χώρες, εμείς θα καταρρύψουμε τους πυράβλους αυτούς και ελπίζουμε πως οι στρατηγικοί μας σύμμαχοι, ΝΑΤΟ, Ευρώπη, στο δικό τους ε, χώρο ασφάλειας θα εξουδετερώσουν απειλές οι οποίες θα στρέφονται όχι κατά των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ αλλά κατά της Ρωσίας. Βεβαίως, οι λεπτομέρειε τέτοιου είδου συνεργασίες χρειάζεται να τις επεξεργαστούμε και μάλλον για πολύ μεγάλο χρόνο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες μας, γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια αχρίαστη σπουδή. Γιατί να πιέζουμε τόσο πολύ. Το Μάρτιο θα γίνει μια συνάντηση των Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ για το θέμα της επιχειρησιακής αντιπυραυλικής άμυνας υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και όπου εκεί κάποια θέματα θα συμφωνηθούν. Εμείς στη Λισαβόνα, ε, αν έχουμε καταλάβει καλά, συμφωνήσαμε όταν τον Ιούνιο συναντηθούν οι Υπουργοί Αμήνης ε, ΝΑΤΟ και Ρωσίας να έρθουμε σε επαφή και με τους εμπειρογνώμονες για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Δεν θα θέλαμε για μια φορά ακόμα να μας φέρετε πρώτε τελεσμένο γεγονότων, γιατί δεν θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε απλώ μια επιχειρησιακή αντιπυραυλική ε, άμυνα του ΝΑΤΟ και να μας πίνε, πείτε αυτή είναι, θέλετε να συμμετέχετε. Δεν νομίζουμε πως κάτι τέτοιο χρειάζεται. Εμείς θεωρούμε πως εάν συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε, θα πρέπει να συγχρονιστούμε και να ακολουθήσουμε το ίδιο χρονοδιάγραμμα συνεργασίας. Εγώ ε, συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και του, προ... και του προτείναμε στις 8 Δεκεμβρίου που είναι η επόμενη συνάντηση ΝΑΤΟ ε, Ρωσίας να παρουσιάσει ένα σχέδιο υλοποίηση των συμφωνηθέντων στην Λισαβόνα και να συναντηθούν και οι εμπειρογνώμονές μας για να συμφωνήσουν πώς θα, ποια μορφή θα μπορούσε να έχει αυτή η επιχειρησιακή αντιπυραυλική άμυνα σε όλες τις περιμέτρους της παραμέτρους της, με συγχωρείτε, έτσι ώστε από εκεί να προχωρήσουμε. Αφήστε με να κάνω και μια προσωπική παρατήρηση. Πιστεύω πως η αντιπυραυλική άμυνα δεν είναι η στρατιωτική απόκριση σε μια πραγματική στρατιωτική απειλή. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα σχέδιο που βασίζεται σε ιδεολογικά σχήματα και που έχει ως σκοπό να ενισχύσει την αλληλεγγύη μέσα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο κοινό project, έτσι ώστε να δώσει ε, ένα τρόπο ώστε να ενοποιηθούν ε, το στρατιωτικό δυναμικό τα υπόλοιπα 10-15 χρόνια. Εγώ δεν νομίζω ότι αύριο ή μεθαύριο κάποιος θα μας επιτεθεί με πυράβλους. Ειδικά ε, μια που έχουμε αυτή τη δυνατότητα με τους ανεχητιστικούς πυράβλους. Πρέπει να σας πω πως μέχρι σήμερα δεν έχει χρειαστεί ποτέ να αναχαιτήσουμε κάποιον επιθετικό πύραυλο και είναι δύσκολο να, φανεί, να φανταστεί κανείς πως οι εχθροί της Ευρώπης θα επιτεθούν εκεί που τους περιμένουν. Ξέρετε πως οι όσοι επιτίθονται συνήθως είναι δειλοί ε, και βρίσκουν τα δύναμα σημεία εναντίον των οποίων κάνουν τις επιθέσεις τους. Το τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι πως δεν νομίζω πως το σύστημα αυτό ε, είναι πραγματικά ε, αξιόπιστο γιατί η επιχειρησιακή αντιπεριβλική άμυνα χρησιμεύει μόνο σε επίθεση μαζικής πυραυλικής επίθεσης. Διαφορετικά δεν μπορείς καν να τη δοκιμάσεις και δεν έχεις μια εξασφάλιση 100% πως μπορεί να αντιμετωπίσει, να καταρρύψει στην πραγματικότητα επιθετικούς πυράβλους. Νομίζω λοιπόν και είμαι πεπισμένο γι' αυτό πως είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε κάποια ιδεολογικά εφευρήματα. Βεβαίως, είναι δική σας απόφαση. Εμείς δεν θα θέλαμε αυτή η αντιπυραυλική άμυνα, αυτή που συζητάμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, να αποτελέσει σημείο διχόνοιας για εμάς. Ε, εμείς θα συμμετέχουμε, παρόλο που έχουμε αμφιβολίες, γιατί θέλουμε μια εταιρική σχέση, θέλουμε μια στρατηγική σχέση μεταξύ ημών, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ε, αντιμετωπίζουμε φαντάσματα απειλών και όχι πραγματικές απειλές. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ε, μπορούμε όμως να συνεργαστούμε. Και βέβαια, νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε άλλες πιο σημαντικές απειλές στην, στο πυρηνικό μας δυναμικό. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών αμυντικών. Είναι εξίσου αρνητικός, ε, αρνητική η κούρσα αυτή με την κούρσα των επιθετικών εξοπλισμών. Α, ξέρετε τι συμβαίνει από το παρελθόν. Όλοι εξοπλιζόμαστε και με τον τρόπο αυτό προκαλούμε ο ένας τον άλλο. Οι δικοί σου εξοπλισμοί οδηγούν στους δικούς μου εξοπλισμούς. Πρέπει λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ε, αποκρίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που πραγματικά αντιμετωπίζουμε για να μην στραφούν όλα αυτά εναντίον μας και να εξασφαλίσουμε το μέγιστο βαθμό ασφάλειας. Ευχαριστώ. ακούτε κάτι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε και στο κοινοβουλευτικό σας παρελθόν. Ε, καμιά φορά πραγματικά ε, είναι ενδιαφέρον αυτό, για το, αυτό που είπατε για τη διπλωματική γλώσσα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας γιατί τονίσατε το θέμα της αξιολόγησης τη απειλή. και την εξέλιξη τη χρονική Υπάρχει μια διαφορετική άποψη. Τα, τους λόγους που και δεν τους βλέπουμε με τα ίδια μάτια μου φαίνεται. Διάφοροι συνάδελφοι έχουν ζητήσει βέβαια το λόγο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Κάμπελ Μπέρμαν που ήθελε και προηγουμένως το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας συγχαίρω που οργανώσατε αυτή την εξαιρετική συνεδρίαση με τόσο σημαντικούς συμμετέχοντες. Το πρώτο μου ερώτημα προς τον κύριο Μπέλ αφορά τη χρήση των πυράβλων αυτών. Θεωρείτε ότι το Ιράν αποτελεί τη βασική απειλή, την υπαρθμόν ένα απειλή στην Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείε όσον αφορά την εκτόξευση πυράβλων. Και κατόπιν των Wikileaks ε, και το τι εξέθεσαν δυστυχώς, αυτό το θέμα της αντιπυραυλικής άμυνας αποτελεί εναλλακτική λύση της ε, στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν που απέτησαν τα κράτη της Μέσης Ανατολής και που αναμένει το Ισραήλ. Δηλαδή, μήπω πρόκειται για κάποια πολιτική αντισταθμιση μια εναλλακτική λύση ε, του να στραφούμε απευθείας κατά του Ιράν. Δεύτερη ερώτηση αφορά σε αυτά που είπε ο κύριος Πρέσβης. Αυτό το σύστημα πυραυλικής άμυνας είναι σε θέση, έχει τις δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί κατά της Ρωσίας, κατά των ρωσικών πυράβλων. Σας παρακαλώ. Ή μήπως μπορεί, τελικά μπορεί αυτό το μυντικό σύστημα να χρησιμοποιηθεί κατά των ε, ρωσικών πυράβλων ή για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά των ρωσικών πυράβλων. Ο κύριος Πρέσβης ε, αναφέρθηκε στο γιατί να πηγαίνουν να κυνηγάνε οι 28 κυνηγοί λαγούς ε, με τέτοια όπλα ενώ, έχουν όπλα που, ενώ, κρατούν όπλα που ε, αντιμετωπίζουν αρκούδες. Ισχύει αυτό που λέμε ή είναι λάθος η εντύπωση αυτή. Ε, δηλαδή αυτοί οι πύραυλοι στρέφονται κατά πυράβλων που μπορεί να εκτοξεύσει το Ιράν. Ευχαριστώ κύριος Βανμπάλ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής ε, τον ε, πρέσβη της Ρωσίας. Συμφωνώ και εγώ ότι χρειάζεται κανείς την πυραυλική άμυνα αν έχει τον φόβο των εκτόξευσης πυράβλων από ε, κάποια χώρα. Προσωπικά δεν φοβάμαι ότι θα μας εκτοξεύσει πυράβλου η Ρωσία. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια διάθεση ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν είμαι όμως βέβαιος ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το Ιράν πυράβλους και έχει, το έχει κάνει. Αν ε, έχει άλλη άποψη η Ρωσική Ομοσπονδία. Θέλω να ρωτήσω, θεωρείτε ότι η πολιτική του Ιράν αποτελεί απειλή προς την περιοχή και αν είτε αυτό το αντιμετωπίσουμε με πυραυλική άμυνα είτε αλλιώς και αν θεωρείτε ότι το Ιράν αποτελεί απειλή για την περιοχή, πώς θα αντιμετωπιστεί η απειλή αν δεν χρησιμοποιηθεί η πυραυλική άμυνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γιάννιας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ή να υπενθυμίσω καλύτερα στον κύριο Ρογκόζιν πως δεν το είδα αυτό βέβαια στο βιογραφικό σας σημείωμα, αλλά πρέπει να σου πω πως κάποια χρόνια, νομίζω μέχρι τα τέλη του 2004, ε, στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου τότε είχατε κι εσείς έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις και θυμάμαι να έχω συζητήσει με εσά τα θέματα για τις σχέσεις Ρωσίας, όπως ήταν σε εκείνο το χρονικό πλαίσιο, με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και θυμάμαι ε, τις που κάνετε για τις σχέσεις της Ρωσίας με το δυτικό κόσμο. Πρέπει να σας πω πως τα 8 χρόνια που πέρασαν η εξέλιξη ήταν πολύ θετική. Τουλάχιστον στην απόκτηση εμπιστοσύνης ε, και στην υπέρβαση ε, δισταγμών και καχυποψίας αμοιβαία καχυποψία. Ποιο θα το φανταζόταν μερικά χρόνια πριν πω θα μπορούσε να γίνει η συνάντηση που κάνουμε σήμερα και θα ήσασταν εσεί εδώ να λάβετε το λόγο και θα ήμασταν κι εμεί εδώ να σα κάνουμε ερωτήσει. Άρα λοιπόν έχουμε προχωρήσει. Θυμάμαι πω το 1998 σε ένα δείπνο που έγινε με τον Χαβιέ Σολάνα εδώ στι Βρυξέλλε που ήταν Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, εγώ είχα κάνει μια ερώτηση, η οποία ήταν προκλητική, ίσως και αφελής. Και σας είπα γιατί δεν σκέφτεστε να ζητήσετε να γίνετε μέλος του ΝΑΤΟ. Εσείς, η Ρωσία. Έχουν περάσει λοιπόν πολλά χρόνια από τότε, γιατί τότε μου είχατε πει, δεν ξέρω αν πρέπει να μπει η Ρωσία στο ΝΑΤΟ ή το ΝΑΤΟ στη Ρωσία. Και αυτό επειδή σας είχε φανεί εξαιρετικά απίθανο να συμβεί αυτό. Και μέχρι τη Λισαβόνα διανύσαμε μια τεράστια περίοδο επαφών και αλλαγής στάσης, καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης, όπου έχει προσεγγίσει τη Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Τώρα για την παράμετρο της ασφάλειας και για τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπορώ να τα πω με δύο λόγια. Το έχουμε συζητήσει πολύ λίγο στην Ολομέλεια, αλλά το συζητούν πολύ τα μίντια. Μιλάμε για μια εντυπωσιακή αύξηση ε, των εξοπλισμών στην Ασία. Ξέρουμε πως υπάρχουν προβλήματα και είχαμε μάλιστα τα πρόσφατα πολύ επικίνδυνα επεισόδια μεταξύ ε, Βορείου και Νοτία ε, Κορέας, αλλά έχουμε την Ινδία και το Πακιστάν και οι δύο πυρηνικέ δυνάμει, την Κίνα η οποία έχει επίση αυξήσει ε, το στρατιωτικό της δυναμικό, την Ιαπωνία, το σύνολο αυτών των χωρών Μιλάμε για Σιγκαπούρη, Μαλαισία και άλλα κράτη της περιοχής με μια πληθώρα προβλημάτων κυριαρχία ή χιλιάδε νησιά για χιλιαδε νησιά. Και η Ρωσία αμφίβολα, δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη σε αυτά τα προβλήματα, νομίζω πως αυτό δεν είναι εκτός των συζητήσεων που κάνουμε σήμερα και θα ήθελα να σχολιάσετε το θέμα αυτό. Και θα κλείσω λέγοντας πως σχολιάστηκε πολύ, ε, ήδη εδώ και κάποια χρόνια, και ακόμα είναι στην επικαιρότητα το κατά πόσο η Ρωσία είναι υπέρ ή βάζει βέτο στην είσοδο νέων χωρών στο, στη συμμαχία. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στην Ουκρανία και τη Γεωργία. Θα ήθελα να σχολιάσετε και αυτό. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν ζητήσει ακόμα τέσσερις συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να είστε, αρκετά, να είστε παρκώς σύντομοι στις ερωτήσει που κάνετε, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να απαντήσουμε. Κύριο Σπιτικό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω πώς ακριβώς ε, μπορεί να περιγράψει κανένα στην ένταξη Ρωσίας μέσα στα πλαίσια της αυτές. Αναφέρθηκε εκείνη η ανάλυση των απατών των, των απειλών, ε, την ανάλυση μιας κοινή ε, ε, αντιμετώπισης. Ε, ακούσαμε προηγουμένως, αλλά αν κατάλαβα τον πρέσβη κ. Ρογκοζίνη, είχα την εντύπωση ότι ήταν παράλληλες εργασίες. Αναλύει δηλαδή η Ρωσία, αναλύει το ΝΑΤΟ. Πόσο έντονη είναι η συνεργασία. Δεύτερη ερώτηση. Κατά πόσον έχει ήδη αποφασιστεί η δομή αποφάσεων, η διακυβέρνηση αν θέλετε αυτού του συστήματος. Και τρίτο, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο πρέσβης κ. Ρογκόζιν που είπε λίγο πολύ, ότι αυτό είναι ένα ιδεολογικό σχέδιο, ένα, ένα σχέδιο που αναφέρεται στην κοινή ασφάλεια, δημιουργία αν θέλετε μια κοινή ασφάλειας. Έτσι το κατάλαβα κύριε πρέσβη τουλάχιστον. Εγώ μόλις ε, τώρα διάβασα μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες μέρες από το Ινστιτούτο για την Έρευνα της Ειρήνης και την ε, Πολιτική Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του, του Αμβούργου. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι το εξής το βάσιμο της πυραυλικής άμυνας δεν θα μπορέσει ποτέ να εξασφαλιστεί τόσο που να μπορούν οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί να βασίζονται 100% σε αυτό. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η υπερατήρηση. Δηλαδή πόση ασφάλεια μπορούμε να πετύχουμε με αυτού του είδους τα ε, σχέδια. Μια ερώτηση για τους δύο πρέσβες που μίλησαν. Ευχαριστώ κύριε Νικολάη. Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πρώτον, πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα, τι γνώμη έχουν οι τι γνώμη έχει ο προσκεκλημένος μας επ' αυτού ή οι προσκεκλημένοι μας, δηλαδή βρισκόμαστε ενώπιον κάποιου κινδύνου αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτά που συζητήθηκαν σήμερα. Και ποια είναι η άποψή σας για την ανάγκη που υπάρχει ελέγχου των εξοπλισμών και των κλασικών αλλά και των πυρηνικών όπλων. Πώς μπορεί το ΝΑΤΟ και η Ρωσία να φροντίσουν να είναι πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος των ε, παραδοσιακών όπλων. Ευχαριστώ. Κύριος Κοράλ. Dziękuję. Dziękuję bardzo. E, panie ambasadorze. Κύριε Πρέσβη, αναφερθήκατε στην ανάπτυξη αμυντικών εγκαταστάσεων στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη και ότι αυτό θα ε, διαταράξει την ισορροπία ασφαλείας. Σε ποια ακριβώς ισορροπία ασφαλές αναφέρεστε, νομική ή άλλη βάση υπάρχει γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτό που μάλλον μου έκλεψε την ερώτηση ο κύριος Μπούτικοφ προηγουμένως. Ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω. Μέχρι ποιο σημείου αναμένετε να εμπλακεί η Ρωσία. Θέλετε να συμμετέχετε στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του συστήματος ε, πυραυλικής άμυνας. Και θέλω και να επιβεβαιώσω αυτό που μόλις είπατε για τα ιδεολογικά ε, προγράμματα στις σχέσεις μας με τη Ρωσία, με την ε, Ένωση, με τον ΝΑΤΟ, με τη Δύση. Ιδεολογικά, φυσικά, επηρεάζουν όλα αυτά τις σχέσεις οι σχέσεις μάλλον επηρεάζονται από τις ιδεολογίε, Αλλά σύμφωνα με αυτά τα οποία διάβασα στο βιογραφικό σας, εσείς είστε ο πλέον κατάλληλος να μιλήσετε για όλα αυτά. Από τη... Για μας ε, η ιδεολογία δεν αφορά την ε, στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία ή ενδεχομένως μια νέα σχέση τύπου ψυχρού πολέμου, αλλά η μελλοντική εξέλιξη της ρωσικής κοινωνίας. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε τη ρωσική κοινωνία να εξελίσσεται προς μια κατεύθυνση στην οποία θα αναγνωρίζουμε παρόμοιες αξίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου, της ελευθερίας ε, σκέψης, τύπου κλπ. Δηλαδή, η συνεδρίαση αυτή επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο το γεγονός ότι οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνη. Το σύστημα πυραυλικής άμυνας μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό στοιχείο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνη και τότε θα αξίζει τα λεφτά του. Ιδάλλως ε, θα είναι μόνο λόγια και δεν μ' αρέσουν αυτά τα λόγια, δεν μ' αρέσουν οι διακηρύξεις που δεν έχουν ουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τέλος η κυρία Γκομές εν συντομία παρακαλώ. Κύριε Πρέσβη, και εγώ αλλά και όλοι διαπιστώσαμε ότι στέκεστε με σκεπτικισμό απέναντι σε αυτό το πυραυλικό σύστημα. Όχι μόνο αναλύοντας την απειλή, αλλά και σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της απόκρισης. Ιδιαιτέρως δε στέκεστε με σκεπτικισμό απέναντι στο αν είναι ο, το Ιράν πηγή βασικής απειλής. Το θεωρείτε αντιπαραγωγικό και στην ουσία λέτε ότι προκαλούμε μόνοι μας αυτό που θα συμβεί. Παρά τα αυτά, συμφωνείτε γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρείτε ότι ελέγχετε ή παρακολουθείτε τι κάνει το ΝΑΤΟ και άρα μπορείτε να το επηρεάσετε. Επηρεάζετε τυχόν εξελίξει από πλευρά ΝΑΤΟ. Ή επίσης, επειδή όντως συμφωνείτε ότι τέτοιες απειλές υπάρχουν. Και είπατε, υπάρχει μια, ένας κατάλογος απειλών. Όλοι λένε για το Ιράν, ε, παρότι δεν έχει θεωρηθεί δημοσίως, αν, ε, αν ονοματιστεί δημοσίως το Ιράν ως ε, απειλή. Υπάρχουν άλλες πηγές, ε, ε, απειλές και κατά την άποψη της Ρωσίας ποιες είναι συγκεκριμένα. Θεωρείτε ότι η Ινδία και το Πακιστάν αποτελούν ίσως σοβαρότερη απειλή όχι μόνο για τα ρωσικά συμφέροντα αλλά τα γενικότερα συμφέροντα της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη και θα δώσω το λόγο και στον κύριο Μπέλ στη διάρκεια της συζήτησης γιατί ετέθη μια ερώτηση στην αρχή προς εκείνον. Νομίζω πως η πρώτη ερώτηση έτσι κι αλλιώς και στον κύριο Μπέλ ε, για το διαμέτρημα αυτών των τουφεκιών που κουβαλάνε οι θηρευτές στο δάσος για την Αρκούδα. Πρέπει να σας πω πως είναι πολύ δύσκολο με όπλο μεγάλου διαμετρήματος να πάει κανείς να κυνηγήσει λαγό. Γιατί δεν θα μείνει λαγός για λαγό στο δάσος. Γι' αυτό εγώ θα σας έλεγα να πάρετε άλλη καραμπίνα μαζί. Εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση αυτή για μας είναι πολύ σημαντική. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε σε συγκεκριμένους χώρους όπου συμπίπτουν τα συμφέροντά μας. Αυτή είναι μια ρεαλιστική συνεργασία. Όμως, πολύ στη Ρωσία και είμαι ειλικρινής, χωρίς διπλωματία σας το λέω, πιστεύουν πως το Ιράν είναι πρόφαση. προφάσει σε αναμαρτίες για να στηθεί μια αντιπυραυλική ομπρέλα για να κυνηγήσουν λαγούς οι δυτικοί. Ίσως αυτές οι φοβίες να μην δικαιολογούνται, ίσως να ανησυχούμε άδικα, μας το λένε οι Αμερικάνοι, πως η αντιπυραυλική άμυνα δεν στρέφεται κατά της Ρωσίας. Ε, εντάξει. Αλλά μετά τον Κορμπατσόφ εμείς πια στα λόγια δεν πιστεύουμε. Εμείς θεωρούμε πως είναι καλύτερο να έχουμε να αποδεικνύουμε με τεκμήρια πως δεν στρέφεται εναντίον μας ε, παρά να μας ε, καλύπτονται με κάποια ωραία λόγια. Εμείς αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στη συνεργασία. Όχι όμως υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια της χώρας μας. Αυτή είναι η λογική που μας διέπει. Γι' αυτό θέλουμε να πείσουμε τους ομολόγους μας στο ΝΑΤΟ πως το σύστημα αυτό θα πρέπει να επικεντρώνεται και τεχνικά και γεωγραφικά και ποιοτικά και χρηματικά να στρέφεται εναντίον των πραγματικών προκλήσεων, των ενδεχόμενων απειλών που αντιμετωπίζουμε, των πραγματικών επαναλαμβάνω. Δεύτερον, και ίσως γι' αυτό δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα, αλλά το σύστημα αυτό της αναχέτησης πυράβλων είναι ένα σύστημα καθολικό γιατί δεν είναι μόνο διαστημικοί, αλλά μπορεί να εκτοξεύονται και από υποβρύχια. Και μπορούν να φέρουν όλων των ειδών της κεφαλές, επίσης μπορούν να εκτοξεύονται και από υπόγειες στοές. Στη θεωρία λοιπόν το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί για να πλήξει στόχους του αντιπάλου μικρού μεγέθους, δηλαδή ένας τέτοιος πύραυλος μπορεί να επιτεθεί σε, ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση και δεν τη βρίσκει κανείς. Άρα λοιπόν θα πρέπει και αυτούς τους παράγοντες να τους λάβουμε υπόψη όταν μιλάμε για έλεγχο των, των συμβατικών ε, όπλων στην Ευρώπη. Για το Ιράν τώρα θα ήθελα να απαντήσω. Ούτε εμάς μας αρέσει και δεν μπορεί να μας αρέσει όταν κάποια χώρα προσπαθεί να αποκτήσει τεχνολογία για όπλα μαζικής καταστροφής. Το έχουμε πει, το είπε και ο κύριος Μπέλ. Η Ρωσική Ομοσπονδία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει στηρίξει μία σειρά ψηφίσματα ε, που προσπαθούν να πείσουν ε, το Ιράν, πως έχει βέβαια τα πραγματικά θεμελιώδη δικαιώματα εξασφάλισης εθνικής του ασφάλειας, αλλά δεν μπορεί να ε, αποκτήσει τέτοια όπλα. Εμείς πρέπει να σας πω ότι γεωγραφικά είμαστε πιο κοντά στο Ιράν από ότι όλοι οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κάποια απειλή, αν υπάρχει κάποιος τρόπος επίθεσης που να έχει αποκτήσει το Ιράν, θα φανεί στη Μέση Ανατολή. Αλλά θα φανεί και κοντά στα δικά μας σύνορα. Για την ασφάλεια, λοιπόν, της χώρας μας αντιμετωπίζουμε το Ιράν με κάθε σοβαρότητα και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την διεθνή κοινότητα έτσι ώστε να διατηρηθεί το σύστημα αυτό μη διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής έτσι ώστε να μην υπάρχει τόσο πειρασμός να αποκτήσουν όλοι τέτοιου είδους όπλα. Όταν λοιπόν συμμετέχουμε στις ομάδες για την αποφυγή της διασποράς και συζητάμε με τους συναδέλφους μας, λέμε για ποιο λόγο εσείς συζητάτε μόνο για το Ιράν. Ας πούμε για όλους. Ποιες είναι οι χώρες. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν αποκτήσει τέτοια όπλα μαζικής ε, καταστροφής. Να τις κατονομάσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνουν μια προσπάθεια συλλογής τέτοιων είδων και απόκτησης ε, τέτοιων όπλων και δεν το κρύβουν. Γιατί λοιπόν δαιμονοποιούμε μόνο μία χώρα. Μήπως πρόκειται εδώ και πάλι για μία ιδεολογική προσέγγιση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις χώρες οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν τέτοιου είδους όπλα. Και δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε αμφιβολίες για το θέμα αυτό. Νομίζω κάποιος από τη Γαλλία βρίσκεται στην αίθουσα, η οποία Γαλλία έχει και αυτή τη δική της θέση στην ομάδα για την αποτροπή της διασποράς ε, των όπλων μαζικής ε, καταστροφής και υπάρχουν πολύ σοβαροί στρατηγοί από τη Γαλλία που θεωρούν ο καλύτερος τρόπος για να εξουδετερώσει κανείς τον πυραυλικό κίνδυνο είναι η διατήρηση Ε, η διατήρηση αυτού του πλεονεκτήματος που έχουμε, του περιορισμού της διασποράς αυτών των όπλων. Και νομίζω ότι η Γαλλία είναι μια από αυτές τις χώρες που θα μας βοηθήσει σε αυτό. Βεβαίως, έχουν τη δική τους προσέγγιση και άλλα κράτη, όπως η Τουρκία που βρίσκεται δίπλα στο Ιράν. Που δεν μπορώ να πω ότι είναι ενθουσιασμένη από το γεγονό πω αυτή τη στιγμή έχει μπει στην κούρσα των εξοπλισμών του Ιράν και προσπαθεί να διαπραγματευτεί και να συνομιλήσει για το θέμα αυτό τη οπλική Απειλή. Εμείς θέλουμε πως ο καλύτερος τρόπος για να διασκεδάσουμε τι ανησυχίε είναι να ζητήσουμε από τη χώρα η οποία προσπαθεί να αποκτήσει κάποιο είδου όπλα για ποιο λόγο το προσπαθεί. Δηλαδή, τι φοβάστε, ποιο νομίζετε πως θα σας επιτεθεί, ποιο σας απειλεί. Μπορούμε να σας δώσουμε εμεί κάποια χέγγια ασφάλεια, έτσι ώστε να μην χρειαστείτε τα όπλα αυτά. Και σας λέω μπορώ να σα πω πως εμείς είμαστε ο μεγαλύτερο υπέρμαχο του πολιτικού διαλόγου και προσπαθούμε όλο το χρόνο και συνέχεια ε, να ε, ξεπεράσουμε τις απειλές που εμφανίζονται. Για το αν θα μπει η Ρωσία στο ΝΑΤΟ, μια άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι δεν είναι επίκαιρο το ερώτημα αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα η Ρωσία, ακόμα και αν ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ, δεν θα μπορούσε. Γιατί στο ΝΑΤΟ υπάρχει μια ομάδα χωρών η οποία μπήκε στο ΝΑΤΟ ακριβώς για να προστατευτεί από τη Ρωσία. Εγώ λοιπόν νομίζω πως αυτή η μία αντικειμενική της φόβη, γιατί εμείς αναφίβολα δεν απειλούμε κανένα και κυρίως στην Ευρώπη που αποτελεί το βασικό μας έχω αλλά καταλαβαίνουμε ότι αντικειμενικά οι χώρες αυτές είναι αλήθεια, φοβούνται. Φοβούνται τη Ρωσία. Και το επαναλαμβάνω, μπήκανε στο Νίκο που λέγεται ΝΑΤΟ, κλείσανε τις πόρτες και φοβούνται πως θα χτυπήσει την πόρτα η αρκούδα που φοβούνται και θα τους πει καλησπέρα. Φοβούνται και οι χώρες αυτές θα μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση ένταξης του Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Το ξέρουμε. Καλά. Αυτή είναι πραγματικά μια δυνατότητα λοιπόν. Και αφετέρου η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θεωρεί πως είναι απαραίτητο για την ίδια. Λόγω της ε, μεγάλης επικράτειας που έχουμε, της μεγάλης γεωγραφικής κάλυψης και δε, δεδομένου ότι δεν έχουμε μόνο σύνορα προς τη Δύση αλλά και προς την Ανατολή, έχουμε την Κίνα η οποία είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εμάς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ε, εμείς βλέπουμε την Κίνα όπως βλέπετε εσείς μερικοί από εσά εμάς. Εάν εμεί λοιπόν μπούμε στην Κίνα, καταλαβαίνετε πώς αυτό θα χειροτερεύσει άμεσα τις σχέσεις μας με τους γείτονε μας προς Ανατολάς. Γιατί βέβαια θα γίνουν σύνορα, σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα, σύνορα του ΝΑΤΟ με την Κίνα. Επίσης, θεωρώ πως αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι να έχουμε εμείς το οπλοστάσιο που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε εμείς τις δικές μας απειλές. Δηλαδή, όπου έχουμε κοινά συμφέροντα θα συνεργαστούμε μαζί σας, όχι μόνο θα στηρίξουμε το διάλογο, αλλά θα μπούμε και σε πραγματική δράση, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε από κοινού τα συμφέροντα των λαών μας και όπου δεν συμπίπτουν τα συμφέροντά μας θα μπούμε σε έναν ειλικρινή διάλογο των προβλημάτων αυτών και θα προσπαθήσουμε μέσω διαλόγου να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Εμάς η συνεργασία μας ικανοποιεί περισσότερο από ό,τι μας ενοχλεί και θέλω να επαναλάβω για μια φορά ακόμα το ΝΑΤΟ δεν είναι ο εχθρός μας. Δεν το θεωρούμε απειλή. Τώρα, σε σχέση με τη Γεωργία και την Ουκρανία, εδώ Έχω μια απάντηση, η οποία δεν εξαρτάται από εμένα, γιατί η Ουκρανία ανεξάρτητα πήρε την απόφαση να στηρίζει μια δέσμευτη πολιτική, δηλαδή να μην μπαίνει σε μπλοκ ούτε ΝΑΤΟ, ούτε οποιαδήποτε άλλη συμμαχία. Μπορώ να σας πω πως το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ κότεψε να διασπάσει στη μέση γεωγραφικά την Ουκρανία και ξέρετε πως όλοι οι πατριώτες στην Ουκρανία θεώρησαν πως καλό είναι το θέμα αυτό να φύγει από την επικαιρότητα. Γιατί ήταν καταστροφικό για την ίδια τη χώρα. Τώρα για τη Γεωργία και εδώ τίθεται το εξή ερώτημα. Δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να δεχτεί μία χώρα που έχει προβλήματα στους κόλπους, που έχει προβλήματα με τις γειτονικέ χώρες. Γιατί ποια είναι τα σύνορα της Γεωργίας. Και προσπαθείτε να λάβετε υπόψη τα λεγόμενά μου. τα παλιά σύνορα της Γεωργίας και τα οποία αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ, τι σημαίνουν. Υπάρχει σύνορο μεταξύ Γεωργίας Απχαζίας, Γεωργίας Νοτίου Ασιτίας. Γιατί τα πραγματικά σύνορα της Γεωργίας σήμερα δεν είναι αυτά με τα οποία παρουσιάζεται για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Ποια αναγνωρίζετε, αυτά που αναγνωρίζει η Ρωσία, γιατί η πραγματικότητα σήμερα σημαίνει ότι υπάρχει Απχαζία, υπάρχει Ασετία και υπάρχει και Γεωργία. Τρία κράτη. Άρα λοιπόν για τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Γεωργίας θα πρέπει να δείτε τι γίνεται ε, με τους εταίρους που, έχουν, που συμβιώνουν με σύμφωνο, πολιτικό σύμφωνο. Δηλαδή η Γεωργία σας βοηθάει στη διέλευση για τα ανατοϊκά οχήματα και τα εφόδια για το Αφγανιστάν. Νομίζω έχει στείλει και κάποια στρατεύματα, δηλαδή είσαστε εταίροι χωρίς να έχετε επισημοποιήσει τη σχέση σας. Είναι μια χώρα ε, που για να γίνει υποψήφιο μέλος θα πρέπει να ε, σέβεται κάποιες ε, παραμέτρους. Τώρα για το κατά πόσο θα κάνουμε κάποιες παράλληλες εργασίες. Ίσως δεν με καταλάβατε καλά. Εμείς δεν είπαμε πως θα γίνουν κάποιες παράλληλες εργασίες για την ανάλυση και τις προκλήσεις που έχει η πυραυλική απειλή. Η ανάλυση που θα κάνουμε του θέματος θα είναι κοινή. Εμείς αυτή τη στιγμή, 8 ε, Δεκεμβρίου, 8 Δεκεμβρίου στη συνάντηση πρεσβευτών στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσία θα λάβουμε απόφαση με ποιο τρόπο θα συσταθεί η ομάδα εμπειρογνωμάων σε αυτό το επίπεδο, μια ομάδα εργασία, ε, η οποία θα έχει έξι μήνε στη διαθεσή τη μέχρι τον Ιούνιο του 2011, έτσι ώστε να συζητήσουν τα διάφορα θέματα, σχηματισμού, φορμάτ κτλ. Θα βρούνε πώ μπορούν το σύστημα αυτό να λειτουργήσει. Δεν θα είναι ένα ενιαίο σύστημα, θα είναι δύο εταιρικά συστήματα τα οποία θα μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό θα οδηγήσει σε ανταλλαγή πληροφοριών για την εκτόξευση, ε, για την αναχέτηση, για τους κινδύνους και πολλές φορές θα ανταλλάξουμε και μυστικές πληροφορίες για τις προοπτικές, ας πούμε, της εξέλιξης αυτών των, της πυραυλικής τεχνολογίας. Μπορεί να ανταλλάξουμε τεχνολογική, τεχνολογικό know-how είτε να προχωρήσουμε σε κάποια βιομηχανική συνεργασία. Μέχρι το σημείο όπου χρειάζεται. Γιατί εμείς θα κάνουμε μια αντιπυραυλική άμυνα η οποία δεν θα απειλεί Αλλήλους, σας είπα, τι κάνουν δύο υπότες που στέκονται πλάτη-πλάτη. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα νότα τους. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε, θα εξασφαλίσουμε ο ένας τον άλλο. Βεβαίως, ε, τα κλειδιά, η είσοδος θα είναι διαφορετική, αλλά θα συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αρχή τη διαδικασία και εγώ αντιμετωπίζω τη διαδικασία αυτή με αισιοδοξία. Πιστεύω ότι σε επίπεδο στρατιωτεχνικό αλλά και πολιτικό υπάρχει η βούληση. Και αν δεν υπάρξει αυτή η βούληση, ε, τότε θα πούμε δεν χάσαμε και τίποτα, τα κλείνουμε και φεύγουμε. Αλλά θα τα πούμε αυτά με ένα διάφορο τρόπο. Για την Κορέα Και βεβαίω ανησυχούμε και εμεί για τι σχέσει που υπάρχουν μεταξύ των δύο κρατών στη χερσόνησο τη Κορέα. Γιατί και εμεί έχουμε εκεί σύνορα στην Άπο Ανατολή. Γνωρίζουμε αρκετά το τι συμβαίνει με τα πυραυλικά προγράμματα τη Βορείου Κορέα. Ξέρουμε πω δεν έχουν ακρίβεια αυτά τα βλήματα, αλλά έχουν μεγάλη εμβέλεια. Μπορούν να φτάσουν μακριά και αυτό μα ανησυχεί. Γι' αυτό λοιπόν τα συγκεκριμένα μέρα για την εξασφάλιση της άμυνάς μας ε, και της ασφάλειας μας στην Άπο Ανατολή έχει, ε, έχουν πάρθει, αλλά δεν καλύπτονται από τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας, γιατί βέβαια η ΝΑΤΟ-Ρωσία καλύπτει θέματα κυρίως ευρωπαϊκά. Ε, θέλουμε η ειρηνευτική διαδικασία στην Κορεατική Χερσόνησο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό. Και θέλουμε να αποφύγουμε την κλιμάκωση αυτών των θερμών επεισοδίων. Τώρα για την πυρηνική ισορροπία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ και πώς αυτό ρυθμίζεται, ξέρετε πώς ρυθμίζεται από την συμφωνία START Ξέρετε πως στη Γενέβη πρόσφατα υπογράφει η νέα συμφωνία, σύμφωνα με την οποία μειώνουμε το επίπεδο στρατηγικής ε, πυρηνικής, ε, πυρηνικών όπλων που έχουμε και μάλιστα ε, οικοδομούμε και περισσότερα μέτρα εμπιστοσύνης, μέτρα ελέγχου και δοκιμής. Εάν λοιπόν μειώνουμε από τη μία το οπλοστάσιό μας, αμοιβαία μειώνεται και η απειλή είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι ήταν κατά τον ψυχρό πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να μην έρθει η αντιπυραυλική άμυνα η οποία όλο και θα αυξάνεται επειδή μειώνονται, ε, μειώνεται ο υπόλοιπο οπλισμό, να έρθει να πάρει το ρόλο που είχε αυτός ο οπλισμός στο παρελθόν. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ισορροπία. Έχουμε την πυρηνική πεντάδα η οποία εμπιστεύεται ε, όλα τα μέρη, άρα λοιπόν εκεί δεν λαμβάνονται καθόλου στρατιωτικο-τεχνολογικά μέτρα που θα διαταράξουν την ισορροπία που έχουμε μεταξύ μας. Ελπίζουμε πάντως ε, πως κάποια μέρα θα επιτύχουμε αυτόν τον κόσμο χωρίς πυρηνικά, που είναι αυτός που επιδιώκουμε. Τώρα, για την αντιπυραυλική άμυνα και για την αναλογικότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μια σύγκριση. και θα ήθελα να γίνει ε, μια σύγκριση με το δηλητήριο των φιδιών. Γιατί σε μικρή ποσότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξει πολύ σημαντικά φάρμακα. Εάν όμως σας δαγκώσει φίδι και είναι πολύ μεγαλύτερο το δηλητήριο που θα λάβετε, μπορεί και να πεθάνετε. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με την αντιπυραυλική άμυνα. Θα πρέπει να προσέξουμε τις αναλογίες, να δούμε ποιος θα, τι ομπρέλα θα έχουμε έτσι ώστε να αποφύγουμε, να καλύψουμε τις μικρής και μέσης εμβέλειας ε, ε, βλήματα, πυράβλους, ε, από χώρες που επιτελούν απειλή. Εάν όμως αρχίζουμε να αναχαιτίζουμε διυπηρωτικούς πυράβλους, έχετε πρόβλημα όχι μόνο με τη Ρωσία, αλλά και με την Κίνα. Και η Κίνα είναι πυρηνική δύναμη και με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί ό,τι συμβαίνει στους δικούς μας κόλπους. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει με ε, μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών με την Κίνα. Αυτό είναι επικίνδυνο και για σας και ιδιαίτερα για μας τη Ρωσία. Είναι ο μεγάλος, τεράστιος, ε, φοβερός γείτονά μας, ο οποίος δεν θέλουμε να εξοπλιστεί μέχρι τα δόντια. Τώρα, για τη Ρωσική Ομοσπονδία, να σας πω που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, εμείς θα πρέπει αναμφίβολα, αδιαμφισβήτητα, να οδηγηθούμε σε ένα, ε, το να ζήσουμε υπό, κοινά, ε, αρχές ανθρωπιστικές, ε, οικονομικές στην Ευρώπη. Θα πρέπει και νομίζω ότι προσωπώ και την αντιπολίτευση σε αυτό που ε- ε- ελέγχθη, ότι είμαστε υπέρ όλων των θεμελιωδών ελευθεριών. Ε, θα πρέπει ο κόσμος να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, να διαδηλώνει ελεύθερα και νομίζω πως ο Ρώσος Πρόεδρος ήταν πολύ ξεκάθαρος όταν μίλησε για εξυγχρονισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Γιατί βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας αποτελεί τον εταίρο κλειδί για ένα διαφορετικό μέλλον. Θέλουμε να ενωθούμε με την Ευρώπη όσο Μα επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουμε. Στο βαθμό που θα μας επιτρέπεται. Αυτό είναι ο στόχο μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρέβη. Κάπως ε, έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά μας όρια. Είναι σημαντικό όμως βέβαια. Είναι η πρώτη σας παρουσίαση εδώ στην υποεπιτροπή μας και τα θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δύο λόγια ίσως από τον κύριο Μπέλτ, γιατί μια ερώτηση ε, του είχε απευθυνθεί. Δύο λεπτά παρακαλώ να επανέλθουμε στο σημείο του Ιράν, που αφορούσε το Ιράν. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομο, ε, Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής θεωρούν ότι το Ιράν είναι η κύρια απειλή όσον αφορά την ασφάλεια στο ΝΑΤΟ. Αντιπρόεδρος την περασμένη εβδομάδα, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένω, ο αντιπρόεδρο Βάιντεν είπε ότι η απειλή προ τι ε, ενόπλε μα και την χώρα μα είναι πάρα πολύ πραγματική, κυρίω από το Ιράν. Και είναι πραγματικά σημαντικό ότι δεν θέλησαν να, ε, να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Διεθνής Οργάνωσης Πυρηνικής Ενέργειας όσον αφορά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών τους κλπ. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διπλωματική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξέβριση λύσης. Και γι' αυτό το μόνο που θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν, είναι, δεν έχουμε ιδεολογική αντιμετώπιση, αλλά μια προνοητική αντιμετώπιση, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η απειλή αυτή. Η ε, πύραυλοι του Ιράν που υπάρχουν σήμερα μπορούν ήδη να ε, φτάσουν σε στόχους στην Ευρώπη. Και η απάντηση της δικής μας κυβέρνησης αυτή τη στιγμή έχει σαν στόχο να αντιμετωπιστεί ακριβώς αυτός ο κίνδυνος. Αναρωτήθηκε ο κ. Πρέσβης γιατί εμείς παίρνουμε στο δάσος τα όπλα αυτά που είναι πιο ισχυρά από εκείνα που χρειαζόμαστε. Και πάλι λέω, είναι θέμα πρόνοιας όπως θα πούνε και οι φίλοι από την βιομηχανία. Γιατί ε, Ε, χρειάζεται πάρα πολλούς χρόνους για την ανάπτυξη αυτών των εξοπλισμών. Θα μας το πούνε και οι συνάδελφοι από την βιομηχανία αυτό. Αυτά τα συστήματα ε, έχει λεχθεί ότι θα έχουν αναπτυχθεί μέχρι το 2010 και όπως σας λέω, οι προοπτικές οι χρονικές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τα συστήματα που θα παρουσιαστούν από τη ΣΥΠΑ σαν συμβολή στην δομή αυτή που θέλει το ΝΑΤΟ δεν ε, είναι δυνατό να απειλήσει την Ρωσία να μην αποδυναμώσει κατά οποιοδήποτε τρόπο την ασφαλή σχέσεις που έχουν οι ΙΠΑ με τη Ρωσία. Και αυτό δεν αφορά μόνο την τοποθέτηση την, ε, των ε, εξοπλισμών αυτών, την τοποθεσία στην οποία έχουν δηλαδή ε, εγκατασταθεί, αλλά και τον τύπο αυτών των αναχειριστών. Μάλιστα, αν θελήσει κάποιος να χρησιμοποιήσει ένας από αυτούς τους αναχαιριστές για να καταρρύψει ένα ICBM που αποστέλνουν οι Ρώσοι προς τη, στη Βόρεια Αμερική, αυτός ο θα κυνηγάει το ICBM χωρίς να το φτάσει ποτέ. Λοιπόν, αν φανταστείτε ας πούμε ότι έχουμε κάποια ε, πλοία τα οποία είναι σήμερα κάπου και ξαφνικά η ΕΠΑ αποφασίσει να βάλει όλους τους, τους τα πλοία στην, στο Βερίγγιο παθμό, και βλέπουμε μετά να περάσουν 10 χρόνια, κατά πόσον υπάρχει μια ιδέα υποθετικού δυναμικού, μπορεί κανένας να κατασκευάσει ένα σωρό σενάριο στο μυαλό του. Στην πραγματικότητα όμως, αυτά τα σενάρια δεν είναι λογικά μεν, και εκτός αυτού ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των 10 ετών αυτών συνεργαζόμενοι με τη Ρωσία θα έχουμε μια νέα σχέση με μια πραγματική στρατηγική σχέση με τη Ρωσία, άρα το σενάριο αυτό θα είναι ακόμα πιο παράλογο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τους διακεκριμένους μας ε, Έχουμε κάποια καθυστέρηση, θα περάσουμε στο τρίτο πάνελ. Κύριε Ζάντρα και που παρακαλώ να περάσουμε εδώ.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

Alors. Hmm? Bien, pardon cette interruption et pardon pour le, le... Λοιπόν, ε, μετά τη διακοπή αυτή και συγγνώμη για την καθυστέρηση, τρίτο πάνελ. Έχουμε τον κύριο Σάντρα εδώ μαζί μας και τον Καμίλ Γκρό, που είναι διευθυντή ε, του Ιδρύματο για την Στρατηγική Έρευνα στο Παρίσι και που ήταν παρόν στην ομάδα εργασία στη Μαδρέν Ομπρέ, που ήταν ε, για το θέμα της στρατηγικής του, ΝΑΤΟ. Ποιος θα το λόγο. Well, first let me thank the... Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνα. για την οργάνωση αυτού του σεμιναρίου, τη ακρόαση τέλο πάντων και την δυνατότητα που δίνεται να μιλήσω. Διάβασα προσφάτα τα πρακτικά της ε, κοινοβουλευτικής ακρόασης που έλαβε χώρα στην Γαλλική Γερουσία πριν από μερικούς μήνες. Πολύ καλή ακρόαση ήταν αυτή και εκεί ακούστηκαν κάποιες ανησυχίες ε, για το ότι δεν υπήρχε ευρωπαϊκή συζήτηση για το θέμα της ε, πυραυλικής άμυνας και χαίρομαι που από τη φυρία έχουμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση. Πολλά ελέγχθησαν ήδη την περασμένη φορά και στα πάνελ που προηγήθηκαν και δεν θα αναπτύξω το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στα δύο βήματα στα οποία συζητήθηκαν τα θέματα της ε, περιοδικής άμυνας στη Λισαβόνα, ένα στα πλαίσια ΝΑΤΟ και το άλλο μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, του Συμβουλίου αυτού. Καταρχήν, όσον αφορά τον ΝΑΤΟ. Η δάση κορυφή τη Λισαβόνα ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για το ΝΑΤΟ, γιατί οι αρχικοί της κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να αναπτύσσουν ένα σύστημα υπεραυλικής άμυνας για να προστατευτούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ΝΑΤΟ, επικράτες και οι δυνάμεις τους. Γιατί λέω ότι ήταν ορόσημο, γιατί αν κανείς διαβάσει το ανακοινωθέν του τηλεφώνου στο προσμένο τους, θα δει ότι εκεί αναφέρεται στην προετοιμασία μια έκθεση για αυτή εδώ τώρα τη διάσκεψη που έλεγε για μελέτη την επόμενη φορά. Περάσαμε λοιπόν από τη μελέτη στην απόφαση. Εγώ πρόσφατα έγραψα ένα άρθρο όπου ακριβώς αναρωτήθηκα κατά πόσον στην Λισαβόνα θα μελετηθεί το θέμα ή θα αποφασιστεί. Το είχα γράψει από το άρθρο πριν από τη Λισαβόνα προφανώ. Και τελικά είδαμε ότι ήταν θέμα απόφαση. Ελήφθη μια απόφαση. Η θα αποφασιστει το ειχα γραψει το αρθρο πριν απο τη λισαβονα προφανω πρόταση στην ε, δεύτερη παράγραφο της δήλωσης ε, της Διάστασης Κορυφή της Αβώνας, για να είναι πληρής πρέπει να αναφέρουμε και το δεύτερο τμήμα, που αναφέρει η απόφαση να κληθεί η Ρωσία να συνεργαστεί μαζί μας. Πάλι, με δύο λόγια αναφέρεται η απόφαση να υπάρχει ε, ανάπτυξη ενός δυναμικού ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα να κληθεί η Ρωσία να συνεργαστεί. Αυτό νομίζω πολιτικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι οι δύο αυτές σημαντικές αποφάσεις αναφέρονται στο ίδιο έγγραφο με απλά λόγια. Τώρα, να αφορά τους στόχους και τις φιλοδοξίες του νέου προγράμματος, αναφέρεται στην παράγραφο 36 της δήλωσης, γιατί διαπραγματευτήκαμε πραγματικά μέχρι μετά τα μεσάνυχτα το έγγραφο αυτό, έχοντας εργαστεί πολλές εβδομάδες προηγουμένως. Λέει εδώ πέρα θα πρέπει η πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ να προσφέρει πλήρη κάλυψη και προστασία για το όλους τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, επικράτη και δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατά της αυξηνόμενης απειλής. Πλήρη κάλυψη. Είναι ο μακροπράθεσμος στόχος. Οι σύμμαχοι όμως αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια σπίδα από τη μια μέρα στην άλλη που να καλύπτει κάθε τετραγωνικό της ε, επικράτειας του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι αδυνάτον από τη μια στιγμή στην άλλη να επιτευχθεί. Γι' αυτό το σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί σταδιακά και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και τις, τους περιορισμούς που μας επιβάλλει η πραγματικότητα αυτή, όπως παραδείγματο χάρη το επίπεδο απειλής, ε, το κόστος και το τεχνικά συγγνώμη δυνατόν. Δεν θέλω να αναπτύξω το LTBMD, αλλά να σας πω ότι υπάρχει βέβαια ένας συσχετισμός ε, με το περιοβλικό σύστημα άμυνας στο ΝΑΤΟ, που είναι η απόφαση να αναπτυχθεί αυτό το πρόγραμμα LTBMD, το οποίο μέχρι στιγμής ε, είχε συγκεντρώσει την προσοχή του στην ανάπτυξη δυνάμεων στο θέατρο πολέμου και τώρα ε, ε, θα μετατραπεί για να μπορέσει να καλύψει και την ευρωπαϊκή επικράτεια. Το LTBMD αυτό πρόγραμμα υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια. Και μέχρι στιγμή είχε σαν στόχο την προστασία από βελιστικού πυράβλου μέχρι 3.000 χιλιόμετρα βεληνικέ. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι η δυνατότητα επικοινωνίας ε, διάταξη και ελέγχου που θα ε, χρηματοδοτηθούν από κοινού. Συζητήθηκε το θέμα 200 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια, όπως είπε ο πρόεδρος Σαρκοζή. Είναι κάτω από τα 200 εκατομμύρια ευρώ για 10 χρόνια. Αλλά αυτά τα χρήματα ε, έχουν σαν στόχο την διεύρυνση του προγράμματος ALTBMD, όχι για το σύνολο του προγράμματος. Το σύνολο του προγράμματος κοστίζει, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά κάτι και για 800 εκατομμύρια. Και πάμε στα 807 εκατομμύρια θα πρέπει να ε, προσθεθούν τα 200 εκατομμύρια για την διεύρυνση ε, του προγράμματος σε γενικές γραμμές. Το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας τώρα. Αυτή η διάσκεψη κορυφής ήταν αποτέλεσμα εντών διπλωματικών προσπαθειών μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων ο Γενικό Γραμματέα Ρασμούστον, η Συμμαχή και η Ρωσία εργάστηκαν σκληρά για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της διάσκεψης κορυφή. Όταν δέχθηκε την πρόταση ο πρόεδρος Μετέγεφ, η πίεση να υπάρχει μια κοινή δήλωση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας αυξήθηκε και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι τελικά πετύχαμε. Ε, η αρχή κρατών και κυβερνήσεων του Συμβουλίου ΝΑΤΟ Ρωσίας ε, ενέκριναν κοινή ε, αναθεώρηση της ε, συμφωνίας για τις απειλές του, του 21ου αιώνα για την κοινή ασφάλεια που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Και συμφώνησαν επίσης για την αξιολόγηση των ε, κοινών ε, κινδύνων από βαλιστικούς ε, πυράβλους. Θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει ακόμα εδώ. Να δούμε κατά πόσο βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Θα πρέπει να σας πω και θυμόμενος πόσο δύσκολο ήταν η συζητήση στο παρελθόν, να σας πω ότι εγώ χαίρομαι να σας πω ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Και γιατί σας το λέω, γιατί ο στόχος στην ανάπτυξη μιας κοινή ανάλυσης απειλής υπάρχει ήδη από το 2002 όταν το Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσίας διδρύθηκε στην Ρώμη Αυτό το έργο αναφέρεται στα κοινά έγγραφα εκεί. Και εγώ είχα αναμειχθεί πριν από μερικά χρόνια στην προετοιμασία ενός παλιού κειμένου που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Είχε μείνει εκκρεμές αν θέλετε το θέμα. Και γι' αυτό το να δούμε ότι τώρα πετύχαμε να οικογραφούν από όλες τις χώρες στην Λισαβόνα τα έγγραφα της κοινή αυτής ανάλυσης είναι κατά τη γνώμη πάρα πολύ σημαντικό γιατί καταδεικνύει αυτό, όχι μόνο σε μας, αλλά και προς τα έξω, ότι μπορούμε, εν τελευταία ανάλυση, να συνυπογράψουμε κοινά έγγραφα σε αυτό το τόσο λεπτό και ευαίσθητο τομέα. Πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν στο μέλλον. Δεν υπάρχει εμβολία. Αλλά αυτή τη στιγμή, 10 μέρες μετά τη διάσκεψη κορυφής, αξίζει να τονίσουμε ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη Σκέψη κορυφής αυτής στη Λισαβόνα. Τώρα να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Πάλι αναφερόμενο στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσίας και μετά θα αναφερθώ στο άλλο θέμα. Καταρχήν, το Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσίας στη Λισαβόνα ανέθεσε στο επίπεδο των πρέσβεων να αναπτύξει ένα μια πλήρη ανάλυση για το μελλοντικό πλαίσιο της συνεργασίας πυραυλικής άμυνας. Ένα θέμα που αναφέρθηκε ήδη προηγουμένως. Ίσως θα αναρωτιέστε τι σημαίνει να υπάρχει μια κοινή ανάλυση. Για να σας πω την αλήθεια δεν έχουμε ακόμα συζητήσει λεπτομέρειες. Δεν θα σε εκπλήξει αυτό βέβαια. είμαστε πολύ κοντά μόλις έχει γίνει η διάσκεψη αυτή στη Λισαβόνα και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το θέμα σε επίπεδο αρμοδίων. Θα υπάρχουν και άλλες επαφές αυτήν την εβδομάδα ήδη, όπως σας είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου Ρωσίας-ΝΑΤΟ για τους πυράβλους, τους οποίους έχω την τιμή να προεδρεύω. Θα το συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Σε εβδομάδα εργασίας αυτήν την εβδομάδα εγώ θα μπορούσα να φανταστώ το έργο αυτό να συμπεριλαμβάνει κάποιες σκέψεις για ενδεχόμενες δομές, ενδεχό ε, επιπτώσεις, νομικά θέματα και άλλα. Δηλαδή, πολλά από τα θέματα που ήδη συζητήθηκαν μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ πάροδο των ετών. Δεν είναι αυτά μυστικά θέματα, τα θέματα της δομής, των επιτελείων, των ελέγχων κλπ. Αυτή ήταν η βάση για την απόφαση που ελήφθη από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Και θα μπορούσαμε να φανταστούμε παρόμοιε συζητήσει μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσία. στη Λισαβόνα σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Μεντβέγερ, εξέφρασε διάφορες σκέψεις που θα έχουν ίσως επιδράσεις στην βούληση της Ρωσίας να συνεργαστεί στην ε, ε, πυραυλική άμυνα ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Ε, θα πρέπει να τα μελετήσουμε αυτά του επόμενου μήνε, να δούμε τι είναι τη Ρωσία και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα να δούμε πώς προχωρούν. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε έτσι ο ένας προς τον άλλο ή με τα νότα ο ένας προς τον άλλον. Ε, Και θα πρέπει να δούμε να μελετήσουμε το θέμα της βάθος και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε αυτή τη συνεργασία και αυτή την ε, πρόοδο. Εδώ μεταξύ θα πρέπει να προχωρήσουμε στην συνεργασία για το TMD, Theater Missile Defense, και είναι πολύ ενδιαφέρον που ακούσαμε ότι θα συνεχίσουμε εκεί που είχαμε σταματήσει με μερικά χρόνια όσον αφορά το θέμα των επιταλείων, των ε, υπολογιστών κλπ. Δύο λόγια όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την πρόοδο. Δύο συγκεκριμένα θέματα που προέκυψαν από τη Λισαβόνα. Καταρχήν ε, να υπάρχει συνεργασία επιτελική ε, έλεγχος και έλεγχος γενικά μέχρι τον Μάρτιο του 2011 για την πυραυλική άμυνα και δεύτερον να υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης για να εφαρμοστεί ε, για, για το πώς θα εφαρμοστεί η πυραυλική άμυνα και αυτό θα πρέπει να προετοιμαστεί μέχρι το 2011 τον Ιούνιο για τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας. Και τελειώνοντα, όσον αφορά τι διαβουλεύσει, οι διαβουλεύσει ε, στοχεύουν στου ρόλου και τι ευθύνε σε πολιτικό επίπεδο και το θέμα της, του ελέγχου τη ποιότητα αυτό γίνεται σε στρατιωτικό επίπεδο. Όσον αφορά το πρόγραμμα δράση που πρέπει να ετοιμάσουμε μέχρι τον Ιούνιο, θα πρέπει να μελετήσουμε το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή μετά τον Ιούνιο. Ίσως το 2020 Ίσως είναι κάποιος χρονικός ορίζοντας αν θέλετε. Για να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε τους επόμενους ε, μήνες, τα επόμενα έτη. Αναφέρθηκα στο 2020, δεν θα σας ε, εκπλήττει γιατί είναι αυτή η γραμμή που έχει προτείνει η Αμερική. Δεν είναι η δυνατότητα, μια από τις δυνατότητες. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή του ισχύοντος LTBMD προγράμματος, τη διεύθυνσή του και το αμερικανικό EPAA. Όλα αυτά θα πρέπει κάπως να ε, συνενωθούν και να συμπεριληφθούν στα χρονοδιαγράμματα για τις συμπληρωματικές εθελοντικές ε, εθνικές συμβολές. Εδώ θα τελειώσω μου φαίνεται. Και οπωσδήποτε η Λισαβόν, όπως είπε και ο πρόεδρος ε, Σαρκοζή, ήταν μια απόφαση αρχής. Οι λεπτομέρειες για την απόφαση αυτή δεν έχουν αναπτυχθεί. Εγώ είχα εμπλεκεί στην αρχική συζήτηση που οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Υπήρξε μια έκθεση από κάποια επιτροπή πέρα στο Συμβούλιο και αυτή ήταν η βάση πάντως τη απόφαση. Η δική μας έκθεση που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο αναφέρει ότι δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί όλες οι λεπτομέρειες. Λέγεται ότι ο διάβολος βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Ίσως αυτό ισχύει για το μέλλον, αλλά οι πληροφορίες που εδόθηκαν αυτή τη στιγμή θεωρήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων επέρκης για να ληφθεί μια απόφαση για το θέμα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ίσως να ακούσουμε τώρα την επόμενη ομιλία ε, του Καμίλ Γκραν. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την ακρόαση. Οι αποφάσεις της Λισαβόνας, η σειρά αποφάσεων που προέκυψαν από τη Λισαβόνα, όπως έχουν μέχρι τώρα περιγραφεί, αποτελούν μια αλλαγή στη θέση του ΝΑΤΟ. Γιατί στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική απόφαση να δεσμευτούν για μια ε, αντιπυραυλική άμυνα που θα προστατεύει και τους πληθυσμούς και τα εδάφη της συμμαχίας. Το σημαντικό σήμερα είναι να διαρωτηθούμε για το τι μας λέει εμάς αυτή η απόφαση, τι, τι σημαίνει για τους Ευρωπαίους. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επισημάνω και θέλω να κάνω μια επισκόπηση των ε, προηγουμένων ε, ομιλιών είναι το θέμα της ε, απειλής. Όλοι στη Λισαβόνα αναγνώρισαν ότι υπάρχει απειλή της διάδοσης των πυράβλων, ότι είναι μια σοβαρή απειλή απαραίτητα να ληφθεί υπόψη μας. Και δεδομένου ότι και μέσω των Wikileaks έχουμε και ενδιαφέροντα στοιχεία, σημαντικό είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά το, το τι έχουν αποκτήσει οι Ιρανοί από τη Βόρεια Κορέα το θέμα των ε, πυράβλων. Οι Βορειοκορεάτες έχουν ε, κατακτήσει όχι μόνο τους περίφους νοτών, τις πυράβλους ε, μικρού βελινεκούς, αλλά και τους πυράβλους μεγαλύτερου τροβελίνικούς, που απειλούν όχι μόνο το Βερολίνο, αλλά και τη Μόσχα πλέον από το Ιράν. Πρέπει λοιπόν, έχουμε ενταχθεί λοιπόν σε μια σε δαιμονοποίηση του Ιράν. Υπάρχουν ε, οι πύραυλοι και ότι μπορούμε να δεχτούμε κάποια πυλή. Βεβαίως δεν πρόκειται για κάτι που θα συμβεί άμεσα, όμως υπάρχει συνέστηση αυτής της εξέλιξης. Ταυτοχρόνως. Μιλάμε για αύξηση της ε, ακτίνας ε, του βεληνικούς αλλά και αύξηση της ε, δυνατότητας. Δηλαδή, μιλάμε για πυράβλους που κατέχει το Ιράν ε, μικρού ή μεσαίου βεληνικούς, αλλά έχουν δυνατότητα ανάπτυξης που πρέπει να και ε, δυναμικότητα που πρέπει εμείς, στην οποία εμείς πρέπει να μπορούμε να αντιταχθούμε. Και όλα αυτά τα λέω, διότι το θέμα της απειλής πλέον δεν είναι θεωρητικό. Για, μεγάλα, για μεγάλο διάστημα αυτοί που επέκριναν την αντιπυραυλική άμυνα ε, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ, γιατί ασχολούμαι το θέμα εδώ και 15 χρόνια, θεωρούσαν ότι η αντιπυραυλική άμυνα δεν ε, ήταν υπαρ... δεν ανταποκρινόταν σε μια υπαρκτή απειλή. Αυτό πάει, πέρασε. Σήμερα η τεχνολογία έχει αρχίσει να λειτουργεί από τη μία πλευρά και οι Αμερικανοί φίλοι μας οι οποίοι έχουν ε, δαπανίσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα αυτό είδαν κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την ε, δαπάνη και από την άλλη η απειλή υπάρχει, ε, εξελίσσεται και μάλιστα γρήγορα. Και αν δούμε την περίπτωση του Ιράν, αλλά βλέπουμε και άλλες ε, χώρες περιοχής που έχουν βαλιστικές δυνατότητες που μπορούν ε, να απειλήσουν την Ευρώπη κάποια στιγμή, ενδεχομένως η Συρία, η οποία από καιρό ενδιαφέρεται για αυτό το σκέλος υπάρχει Υπάρχουν και υποπεριφερειακές ε, δυνάμεις που όμως μπορεί να εξελιχθούν και μπορεί κανείς ε, ε, όταν ένας γείτονα, ας πούμε το Ισραήλ μπορεί να απειλήσει έναν άλλο γείτονα που όμως είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, ας πούμε την Τουρκία, τότε υπάρχουν θέματα. Σήμερα λοιπόν οι χώρες αυτές δοκιμάζουν, αποκτούν, αναπτύσσουν βαλιστικούς πυράβλους μικρού και μέσου βεληνικούς. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει λοιπόν κανείς να διερωτηθεί αν όλα αυτά τα προγράμματα θα, οριμάσουν και πότε, αν μιλάμε για ένα χρόνο ή για δεκαετία. Εν πάση περιπτώσει τα θέματα είναι δευτερεύοντα όταν σκεφτούμε τι είδους ε, στρατηγικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν, όπως είπαμε και προηγουμένως δηλαδή. Η αποφάσεις για την αντιπυραυλική άμυνα από πλευράς ΝΑΤΟ θα χρειαστούν καμιά δεκαετία για να υλοποιηθούν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Τώρα, όσον αφορά τώρα τη Λισαβόνα, θέλω να, πω, να σας πω μερικές σκέψεις μου για αυτά τα οποία αποφασίστηκαν και αυτά τα οποία δεν αποφασίστηκαν στη Λισαβόνα. Συμφωνώ απόλυτα με ε, το γεγονός ότι ανέλαβε μια πολιτική αποστολή η Λισαβόνα, αλλά δεν θα πρέπει όλες οι συζητήσεις να επικεντρώνονται γύρω από την αντιπυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ. Πρώτον, η αξιολόγηση της απειλής. Και εδώ πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Πρέπει τα μέχρι ότου τα πράγματα γίνουν πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει μια συζήτηση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μέχρι ποιου σημείου πρέπει να ε, αν εντοπίζεται μια συγκεκριμένη απειλή και όπως ξέρετε η Τουρκία αντιτίθεται στην αναφορά στο Ιράν στο πλαίσιο αυτό και υπάρχουν και άλλοι σύμμαχοι που θεωρούν ότι το Ιράν είναι μια ε, υποβόσκουσα απειλή. Και τώρα, το ποια, ποιες φάσεις θα καλύψουμε ε, θα εξαρτηθεί από την πραγματικότητα της απειλής. Δηλαδή οι Αμερικανοί είπαν ότι οι τελευταίες φάσεις, οι τρία και τέσσερα που μόλις ε, σας περιγράφησαν, δεν θα υλοποιηθούν αν η απειλή του ε, Ιράν εξαλειφθεί λόγω ας πούμε διπλωματικών Άρα πιο συγκεκριμένα πρέπει να, να αποφασίσουμε αν πρέπει να μιλάμε ε, για τις ε, απειλές που είναι μικρότερου βεληνικούς ή μεγαλύτερου βεληνικούς. Όλα αυτά πρέπει να διευθετηθούν. Δεύτερο ζήτημα που επίσης συζητήθηκε πολύ εν, καθοδόν προς τη Λισαβόνα, το θέμα της αποτρεπτικότητας σε σχέση με την αποτροπή. Γνωρίζετε ε, ότι έχει τεθεί ένα θέμα αν η αντιπυραυλική άμυνα αποτελεί υποκατάστατο ή συμπλήρωμα της αποτρεπτικής ε, δυνατότητας. Ε, ενισχύει, λέμε, την, την, την ή όπως λέμε στα αγγλικά bolster την δηλαδή το πρόβλημα της απειλής των πυράβλων ε, θα συνεχίσει το ΝΑΤΟ να το αντιμετωπίζει με μια μεικτή δυνατότητα με ε, τα συμβατικά όπλα με τα πυρηνικά όπλα και με την ε, αντιπυραυλική άμυνα και αυτό πιστεύω ότι θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε αυτό το μείγμα όταν συζητάμε το θέμα αυτό και σε άλλους χώρους. Τώρα, τρίτον, η τεχνική του μελλοντικού συστήματος, θα είμαι σύντομος πολλά υπόθηκαν, πρέπει καταρχήν να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο αποφασίστηκε στη Λισαβόνα και αυτό το οποίο... Ε, ε, ετέθη στον προπολογισμό της ε, Λισαβόνας και μας το θύμισε αυτό ο Ρομπέρτο είναι αναπόδραστο στοιχείο του συστήματος ALTBM δηλαδή συστήματος ε, ελέγχου και διοίκησης. Πρόκειται δηλαδή για προσθήκη 200 ή 800 ακόμα εκατομμυρίων σε αυτά που έχουν προϋπολογιστεί, ώστε να υπάρχει ένα δίκτυο, ε, ένα δίκτυο υπολογιστών που να είναι σε θέση να κινητοποιήσει, να συνδέσει τους διάφορες αμερικανικούς κυρίως ε, αισθητήρε που υπάρχουν. Λοιπόν, σε ένα, είμαστε σε μια φάση όπου με 200 εκατομμύρια δολάρια θα ε, προστατεύσουμε την Ευρώπη με ένα βαλιστικό σύστημα πυράβλων, με περισσότερα εκατομμύρια δολάρια, θα επιτρέψουν στους Αμερικανούς ε, και άλλους ίσως στο μέλλον, το παρόν Αμερικανούς, να προστατεύσουν την Ευρώπη απέναντι σε κάποιες βαλιστικές απειλές. Αυτό για να σας κάνω τη σύγκριση Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια των τελευταίων, της τελευταίας δεκαετίας ε, ε, δαπάνησαν 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ε, πυράβλων θεάτρου. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι με 200 εκατομμύρια ευρώ, παρότι η ισοτιμία είναι υπέρ του ευρώ αυτή τη στιγμή, θα μετατρέψουμε κατά ανάγκη την κατάσταση που ισχύει στην Ευρώπη τα μέσα που θα αναπτυχθούν στην Ευρώπη είναι, θα στοιχήσουν ίσως ε, και στον Αμερικανό φορολογούμενο, αλλά εν περιπτώσει θα στοιχήσουν 20-40 δις δολάρια χωρίς τις ενδεχόμενες ε, συμμετοχές από πλευράς Ευρωπαίων που μπορεί να ανεβούν σε πολλά εκατομμύρια ευρώ αν αποφασιστούν αυτά τα προγράμματα. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε όταν συζητάμε για τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, πρέπει να θα μπορέσει ε, το αμερικανικό σύστημα να συνδεθεί με το σύστημα του ΝΑΤΟ. Είναι μια ε, καλοπροαίρετη και φιλική προς το χρήστη ε, ερμηνεία, ίσως είναι λίγο υπερβολική η σύγκριση με το σύστημα που, ένα σύστημα που το συνδέουμε με την τηλεόρασή μας. Σε βάση περιπτώσει, το θέμα εδώ είναι πώς λειτουργεί. Από τη μία με δυνατότητες ε, αισθητήρων και και με την αναχέτηση που την έχουν οι Αμερικανοί και αν όλα τα συστήματα λειτουργούν κατά ακριβώς τον ίδιο τρόπο, αυτά όλα πρέπει να λυθούν και βεβαίως θα διαπιστώσετε ότι οι, ε, αυτά βρίσκονται σε πλοία τα οποία εξορισμού κινούνται, άρα σε ένα πλαίσιο που η βαλιστική απειλή είναι πιο περισσότερο παρούσα ε, στην ε, Ασία ή στη Μέση Ανατολή, ε, οι Αμερικανοί να πούν, απολύτως δικαιολογημένα, ότι αυτές τις δυνατότητες θα τις μετακινήσουμε στις ζώνες όπου ο κίνδυνος είναι πιο πιεστικός. Αυτό είναι ένα θέμα για τους Ευρωπαίους. Τι θα κάνουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι, θα δώσουν ε, τις δυνατότητές τους στους ε, Αμερικανούς, θα αναπτύξουν δικές τους, θα ε, κινηθούν μέσω του ΝΑΤΟ. Το επόμενο θέμα είναι ο μηχανισμός ελέγχου και οι κανόνες εμπλοκής του μελλοντικού συστήματος. Είναι δύσκολο να πούμε κατόπιν όλων αυτών ότι ένα τέτοιο σύστημα που έχει τόσο σύντομους χρόνους απόφασης ε, θα ε, εξαρτηθεί από τις αποφάσεις ενός Αμερικανού ε, ναυάρχου που είναι ο Σακέρ. Γιατί δεν βλέπουμε φυσικά απόφαση του, Συμβουλίου, του Βορειοατλαντικού Συμφωνίου. Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα εδώ και στο σύστημα όπου οι αισθητήρε, οι ταραντάροι, οι δορυφόροι, οι το σύστημα αναχέτησης που μας το παρέχει ένας σύμμαχος, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ποια είναι η ε, αλληλουχία της λήψης αποφάσεων, της διοίκησης. Είναι τεχνικό, αλλά βεβαίως είναι και πολιτικό το ζήτημα αυτό. Και όλα αυτά πρέπει ακόμα ε, να αποφασιστούν, δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Ένα τρίτο τεχνικό ζήτημα. Ποια είναι η προσφορά, η συνεισφορά των άλλων Ευρωπαίων. Υπάρχει εισφορά, συνεισφορά από την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία και πέραν αυτού θέλουν ε, να συνεισφέρουν οι Ευρωπαίοι σε είδος και με ποιο τρόπο. Ας πούμε, ο Ποπέλ είπε, υπάρχουν μέσα, αλλά η συνεισφορά αυτή δεν είναι αποφασιστική για τη λειτουργία του συστήματος. Και σε λίγο θα μιλήσω για το τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη στο θέμα αυτό. Τέλος, συζητήθηκε διαμακρών το θέμα συνεργασίας με τη Ρωσία. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολιτικά ωφέλη από αυτή τη ρύθμιση, είναι απολύτως ευκταία Πρέπει να ησυχάσουμε τους φίλους μας Ρώσους ότι η πυραυλική άμυνα δεν στρέφεται κατά της δυνατότητας της Ρωσίας. Επίσης ε, αφορά τις σκέψη, την αντιμετώπιση από, τη Ρωσία το θέμα, από το θέματος αυτού, που είναι κάτι το πολύ καλό. Τώρα υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα και εδώ πρέπει να κάνουμε κάποια διάκριση αυτό που είναι, μεταξύ αυτού που είναι απολύτω ε, επιθυμητό, όπω είπε και ο κ. Ρογκοζίν, δηλαδή το θέμα τη αξιολόγηση τη απειλή και μια σοβαρή συζήτηση από αυτού για να ε, ε, συγκλίνουν οι αξιολογήσει ΝΑΤΟ και Ρωσία. Ίσως ένα σύστημα προειδοποίηση σχετικά κοινό ή μια κοινή προσέγγιση δύο συνόλων. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε να ωφεληθούμε κοινέ αντιπυραυλικέ ε, δαπάνε, ε, Είναι δύσκολο, είπαμε ότι είναι δύσκολο ήδη να γίνει αυτό ανάμεσα σε 28 συμμάχου. Τώρα, ανάμεσα σε 29 όπου, όπου η άλλη χώρα έχει διαφορετικά πρότυπα και προσεγγίσει ίσω να περιπλέξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει το πιθανότερο είναι να ακολουθήσουν μακροσκελή συζητήσεις χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα και τελικά μπορεί να πούμε ότι θα καταλήξουμε σε δύο χωριστά συστήματα που συνεργάζονται με διαφορετικούς τομείς, γιατί το ρωσικό, η ρωσική πλευρά είπε στα πλαίσια της συζήτησης μετά τη Λισαβόνα, όπως εμφανίστηκαν στο ρωσικό τύπο, ότι, θεωρούν, ότι βλέπουν ένα σύστημα που θα είναι, αποτελείται μάλλον από δύο συστήματα back to back και όχι το ένα δίπλα στο άλλο. Πρέπει να μην μας διαφεύγει αυτό, παρότι πρέπει να χαιρόμαστε που έχει το ΝΑΤΟ την πολιτική θέληση να συνεργαστεί με τη Ρωσία και η Ρωσία επιθυμεί να εμπλακεί σε αυτή τη συνεργασία. Τώρα, εν κατα, ε, κατακλείδη. Θέλω να επανέλθω στη θέση της Ευρώπης στο πλαίσιο αυτό και χαίρομαι που η Υποεπιτροπή έπλεξε να ασχοληθεί με το ζήτημα και ο κύριος Απρά μίλησε για τις ακροάσεις της Γαλλικής Γερουσίας. Είμαι από αυτούς που ανησυχούν από το γεγονός που η... ότι η Ευρώπη δεν το σκέφτεται αυτό το θέμα, δεν συζητήθηκε. Το είπα αυτό. Η Ευρώπη, η η Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαίω, ίσω ε, αποφασιστεί στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, εγώ θεωρώ. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη απέναντι σε αυτό, σε αυτή την κατάσταση. Το πιθανότερο σενάριο είναι να συνεχίσει να μην κάνει τίποτα και να επιλέξει την ε, επιλογή του λαθρεπιβάτη που θα μπορέσει να καλυφθεί ε, το έδαφος του, η Ευρώπη δηλαδή, και να μην ξέρει, να ξέρει όσο τον λιγότερα από αυτού και να επιτρέψει στους Αμερικανούς να ασχοληθούν με το θέμα. Είναι μια λύση που βεβαίως είναι cost effective παρόλο που ε, έχει και την ευφυΐα της παρότι δεν ξέρουμε τι θα συνεπάγεται αυτό σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν. Υπάρχει η, ο, μηχανική, ο τρόπος που θα ε, χτίσει το σύστημα το, το ΝΑΤΟ. Επίσης, η Ευρώπη δεν θα οι Ευρωπαίοι δεν θα εξυπηρετούνται τόσο καλά όσο οι Άπωνες ας πούμε ή οι χώρες του κόλπου γιατί αυτές ε, είχαν ε, την προθυμία να δαπανίσουν κάποια χρήματα. Άρα η Ευρώπη τίθεται σε κάπως ιδιαίτερη ε, κατάσταση και κυρίως δεν θα είναι σε θέση να επηρεάσει την αρχιτεκτονική του νέου συστήματος και να διατυπώσει την άποψή της επ' αυτού. Τώρα, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται στο θέμα της διάδοσης βαλιστικών πυράβλων, κυρίως στο διπλωματικό πεδίο. Είχα και λόγω των σπουδών μου την ευκαιρία να υλοποιήσω μια σχετική απόφαση του Συμβουλίου που επικεντρώνει στο θέμα της διάδοσης ε, μια δραστηριότητα πάρα πολύ χρήσιμη που εκ των υστέρων ε, ασχολείται με το θέμα της διάδοσης των ε, βαλιστικών αλλά που ελάχιστα κάνει για αυτή καθεαυτή την απειλή. Είμαι λοιπόν πολύ υπέρ και το έχω ήδη πει του η European Defense Agency να ασχοληθεί με το θέμα και να ασχοληθεί όχι μόνο με το θέμα της αρχιτονικής αλλά και το θέμα της τεχνολογίας. Δηλαδή αν θέλουν οι Ευρωπαίοι να ασχοληθούν με το ζήτημα, δεν θα πρέπει να ε, ασχοληθούν ε, ε, σε χρόνο που δεν θα είναι ο κατάλληλος. Πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμός με το ΝΑΤΟ και σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να εξελιχθούν προς αυτή την κατεύθυνση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας Βεβαίως, να γίνουν μελέτες που αφορούν ε, τα χρήσιμα τεχνολογικά στοιχεία. Αυτή είναι μια σημαντική ε, συνεισφορά με χαμηλό κόστος που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να κατανοήσουν το ζήτημα και δημοσιονομικά ή να αναπτύξουν, ε, με δημοσιονομικά κατάλληλο τρόπο, να αναπτύξουν κάποια στοιχεία τεχνολογίας. Δεν κάνω τώρα κριτική, δεν επικρίνω τον οργανισμό. Ε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ε, λέω ότι και πέραν ε, ε, ε, αυτού υπάρχουν κάποιες υφιστάμενες συνεργασίες και θα ήταν ενδιαφέρον να μπορέσουν να πτυχθούν αυτές οι συνεργασίες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ με τους οποίους, με τους οποίους οργανισμούς δεν είναι ασυμβίβαστοι. Τώρα, στην ευρωπαϊκή βιομηχανία υπάρχουν κάποιες δυνατότητες. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Ε, μιλάμε για δαπάνη 100 δισεκατομμυρίων στην επόμενη δεκαετία για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάπου στο επίπεδο των Αμερικανών. Όχι. Μιλάμε για κάποιες ε, δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε αυτό το τεχνολογικό ε, αγώνα, να μπούμε και εμείς μέσα σε αυτή την προσπάθεια. να φτάσουμε το ένα δις ας πούμε που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να έχουν τη δυνατότητα να ε, συμμετέχουν, να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια σε ένα διάστημα 10-15 ετών. Όλα αυτά λοιπόν ε, σημαίνουν ότι υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα αισθητήρε είτε στα ε, ραντάρ είτε στους δορυφόρους Υπάρχουν επίσης ε, και υπάρχει τεχνολογία που αναφέρθηκε προηγουμένως, στο πρόγραμμα MEAD και μια σειρά άλλα ε, προγράμματα που δεν είναι θεωρητικά, αλλά που ε, δυστυχώς δεν έχουν χρηματοδοτηθεί επαρκώς για να φτάσουν σε, στη φάση της επίδειξης και να μπορέσουν να, μπουν, να προχωρήσουν έτσι και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας είμαι βέβαιος θα υπενθυμίσουν τι ε, υπάρχει. Και είναι κρίμα που δεν σκεφτόμαστε την ανάλυση της ε, αντιπυραυλικής άμυνας και τους ε, ευρωπαϊκούς περιορισμούς είναι ένα σύστημα που αναπτύσσει το ΝΑΤΟ. Πολύ συχνά ε, έχουμε ένα θέμα με ε, ενός μόνο αντιπάλου, το one-on-one, -on -one, on ενω Ευρώπη, από την Ευρώπη υπάρχουν πολύ πιθανοί στόχοι. Τι θα γίνει ε, αν πρέπει ένα πλοίο να επιλέξει μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών στόχων. Είναι κάτι που εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να το συζητήσουμε, να αναπτύξουμε την τεχνογνωσία μας, ε, τη δυνατότητά μας να συνομιλούμε με τους Αμερικανούς και με τη Ρωσία βεβαίως να, προσφέρουμε λοιπόν και να μην είμαστε απλώς ένας λαθρεπιβάτης σε αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι λοιπόν για μία ακόμα φορά που ε, σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία να το συζητήσουμε το θέμα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ γιατί ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Είχαμε τις πρώτες πολιτικές ε, παρεμβάσεις σήμερα που οδήγησαν σε κάποια σύγχυση. για τα συστήματα και ότι καλύπτουν τα αριθμητικά στοιχεία που υποβλήθησαν και όσον αφορά βέβαια και την προοπτική των εργασιών που πρέπει να γίνουν και στο επίπεδο ΝΑΤΟ και στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εμεί εκφράσαμε τι ανησυχίες μας πλησιάς, που ανέφεραν το θέμα γενικά ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσουν τα θέματα. Έχουμε αρκετή καθυστέρηση. Εγώ δεν έχω ο, ερωτήσει. Κυρία Κόπ, έχει το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και του δύο για τι παρεμβάσει σα. Η ερώτησή μου αφορά την, Τουρκία ε, την διοίκηση των δύο συστημάτων. Ε, είπατε ότι το Ιράν δεν αναφέρεται στην απόφαση του, της Λισαβόνας, ότι όλη η επικράτεια της Ευρώπης θα καλύπτεται από τα συστήματα αυτά και ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση του συστήματος. Τα δύο πρώτα ερωτήματα βρήκαν απάντηση, το τρίτο όμως όχι. Η ερώτηση αυτή για τη διοίκηση θα αρχίσει προσεχώς. Μπορούμε να φανταστούμε ότι οι Αμερικανοί θα προτίθενται να μοιραστούν με άλλους την δίκηση αυτή, γιατί όπως είπε και ο κύριος Γκρόντ, το δυναμικό είναι στο σύνολό του σχεδόν αμερικανικό και δεν ξέρω κατά πόσον οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν δικό τους δυναμικό. Θα μπορούσε δηλαδή να ληφθεί υπόψη κάποια απόφαση για τη δίκηση που δεν θα είναι μόνο αμερικανική. καλό. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει στο ερώτημα αυτό. Ξέρουμε όμως ήδη ότι για διάφορες χώρες, για την Τουρκία, παραδείγματο χάρη που αναφέρθηκε ήδη, και άλλες χώρες, η Γαλλία και άλλες, είπαν ήδη μπλιστάκες ότι το θέμα του ελέγχου και της διοίκησης είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να υποβληθεί κάποιο αποτέλεσμα για τον Μάρτιο ήδη, για την διάσκεψη του Μαρτίου. Εγώ προς το πάντως δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση γιατί υπάρχει ακόμα πολιτική απάντηση για το θέμα αυτό. Καμίγη το κατά θέλει. Ναι, Πράγματι δεν υπάρχει οριστική απάντηση. Μπορώ να σας πω ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιλέξιμες λύσεις. Πραγματική συζήτηση θα ε, αφορά τους κανόνες δέσμευσης. Γιατί θα έχουμε ένα θέμα που θα ζητάτε απόφαση σε δευτερόλεπτα, σε λεφτά. Δεν μπορεί να υπάρχει συζήτηση. Δηλαδή θα αποστελεί ένα πύραυλο από το Ιράν. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα θα αναχαιριστεί, θα αναχαιριστεί ή τι. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει αποστολή. Γιατί ότι όταν ένα πύραυλο προέρχεται από την εξή ε, χώρα προ την αυτή κατεύθυνση, θα ξεκινήσει ο μηχανισμό αναχέτηση με τρει αναχαιριστέ, ανάλογα που θα πάει κλπ. Είναι μια τεχνική συζήτηση αφενός καλύτερη επιλογή δηλαδή να είναι επιτυχή η αναγέννηση και μια πολιτική συζήτηση. Κατά πόσο να αποφασίσουμε ότι ό,τι ξεκινάει από το Ιράν προς την Ευρώπη θα πρέπει να αναγυριστεί. Ακόμα και αν πρόκειται για παράδειγμα χάρη για εκτόξευση δορυφόρου. Ξέρω εγώ κάπως υπερβάλλω αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τεχνικά Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το ένα λέει ότι εντάξει, στο τέλος θα έχει κάποιος ε, τα κλειδιά της δίκησης. Δεν ξέρω αν θα βρίσκεται στην Τουρκία αυτό, θα βρίσκεται όπου δεν ξέρω. Υπάρχουν διάφορες ιδέες. για να υπάρχει ίσω και κάποια δυνατότητα παρακολούθηση του τι γίνεται εκεί και είναι σημαντικό να υπάρχει μια σημαντική θέση στην αλυσίδα αυτή τη διοίκηση. Η τελευταία αναλύση όμω. η απόφαση μπορεί να είναι πολύ κάθετη. Μέσα στα πλαίσια δηλαδή τη θεωρητική διοίκηση του ΝΑΤΟ. Από την άλλη μεριά μπορεί να υπάρχει μια απόφαση πιο ευρύ ε, όσον αφορά το εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει όμω το ευρωπαϊκό το εθνικό δυναμικό. Είναι δύσκολο να πει κάποιο. Εγώ θέλω να έχω το λέγιν για την αναχέτηση όταν δεν υπάρχει κανένα εθνικό δυναμικό. Είναι κάπως υπερβολικό. Παράδειγμα. Συνεργασία Ισραήλ-Αμερικανών για την ε, Ισραηλή ε, άμυνα υπάρχει ένα σύστημα ε, έγκυρης προειδοποίησης ολιγόνιν ε, από το οποίο ωφελούνται οι Ισραηλινοί. Από την άλλη μεριά, η αποφάσει για την ανέχετηση ή όχι πυράβλων που κατευθύνονται προς το Ισραήλ λαμβάνονται από το Ισραήλ. Δεν αναμειγνύονται εκεί οι Αμερικανοί. Είτε πρόκειται για Ισραηλοαμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικών ε, ε, αντιπυραυλικής άμυνας ή για καθαρά Ισραηλινά συστήματα. Όλες οι χώρες που έχουν αντιπυραυλική άμυνα σήμερα, η Ρωσία, το Ισραήλ, η ΙΠΑ έχουν πολύ αυστηρές ε, διοικητικές γραμμές εθνικές και θα πρέπει να δούμε τι, πώς θα λειτουργεί το θέμα σε πολυεθνικό πλαίσιο. Η σύγκριση που κάνω συχνά είναι με τις αποφάσεις αναχέτησης των λεγόμενων πειρατικών αεροπλάνων, renegade όπως τα λέμε. Είναι δύσκολο να ληφθεί η απόφαση να καταληφθεί ένα πολιτικό αεροπλάνο, γιατί υποτίθεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάντως αυτή είναι οπωσδήποτε εκάστοτε εθνική απόφαση πολιτική, μια απόφαση που δεν λαμβάνεται αυτόματα. Δεν λέει υπάρχει κάποιος υπολογιστής που αυτόματα αποφασίζει αυτό το αεροπλάνο θα καταληφθεί επειδή πετάει από εδώ ή από εκεί κλπ. Υπάρχει πάντα μια πολιτική διάσταση που λαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό ή από έναν Υπουργό που έχει, τον οποίο έχει κρυφθεί η ευθύνη αυτή. Και όπως είπαμε, η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μερικά λεφτά. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε αναχέτηση σημαίνει υπάρχει κίνδυνος με τα θράψματα, ε, με τα προβλήματα με τη χώρα από την οποία ξεκίνησε ο πυρόβλος αυτός, πρόκληση ίσως ε, εντάσσεων κλπ. Πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μου να λαμβάνει η απόφαση πολιτικά. Και όχι ο πλήρχος του εν λόγου σκάφους αποφασίζει ότι θα αναχαιτήσει ή όχι πρωτού περάσει ε, στο βιομηχανικό θέμα, έχω μία τελευταία ερώτηση. Δηλαδή, πολιτικά και τεχνολογικά, η διαδικασία στην οποία, με την οποία ξεκινάει το ΝΑΤΟ, κατά τη γνώμη σας, είχε κάποιο αποτρεπτικό αποτέλεσμα στα προγράμματα των χωρών που αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή αυτούς τους εξοπλισμούς. Δηλαδή το γεγονό ότι τεχνολογικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ιδίω από του Αμερικανού, αλλά όχι μόνο, αυτό αποτρέπει κάποιες χώρες να προχωρήσουν σε αυτό το τεχνολογικό άλμα για τα βαλιστικά τους προγράμματα. Η δική μου αξιολόγηση είναι η εξή και είναι διπλή. Καταρχήν, η αντιπυραυλική άμυνα έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα και αποθαρρύνει κάποια κράτη από το να ξεκινήσουν προγράμματα απόκτηση πυράβλων, γιατί το κόστος είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Δηλαδή, για να αποκτήσει κανείς βαλιστικούς πυράβλους, που είναι μία ασύμμετρη απειλή, μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει παρόλο που δεν θα αποκτήσει πλήρες οπλοστάσιο για την μεταφορά για παράδειγμα χημικών ή βιολογικών όπλων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως για να μπει κανείς σε, αυτό τον, σε αυτή την κούρσα εξοπλισμών το κόστος είναι υψηλό και γι' αυτό είναι πολύ σωστό να αποθαρρύνουμε τα κράτη από το να προσπαθούν να αποκτήσουν κάποιο είδους βαλιστικούς πυράβλους, γιατί θα γνωρίζουν ότι μέσω της αντιβαλιστικής άμυνας που θα έχουμε εμείς δεν θα τους επιτρέψουμε να τα χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή το κόστος εισόδου σε αυτό το παιχνίδι να είναι πολύ υψηλό γιατί θα τους εξηγούμε από την αρχή ότι έχουμε μια πολύ καλή δυνατότητα αναχέτησης αυτών των πυράβλων και ότι οι πύραυλοι οι οποίοι θα αποκτήσουν τεχνολογικά δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τη δική μας αντιπυραυλική ασπίδα. Δηλαδή το να έχουμε μια ε, μικρή εμβέλειας βαλιστικό πύραυλο που θα χρησιμοποιηθεί. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τον αναχαιτήσουμε πάντοτε σίγουρα γιατί είναι σαν να κυνηγάει κανείς μια βελόνα που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Όμως, Οι προκλήσεις σήμερα είναι διαφορετικές. Δεν είμαστε στις φάσεις του ψυχρού πολέμου που φοβόταν κανείς μια πυρηνική επίθεση. Μιλάμε για επιθέσεις οι οποίες είναι στοχευμένες, μικρές, αρκετά πρωτόλιες πολλές φορές σε επίπεδο εξοπλισμού και αυτές προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Το θέμα είναι κατά πόσο μια χώρα που είναι ιδιαίτερα αποφασισμένη να παρακάμψει αυτό το σύστημα να το κάνει είτε χρησιμοποιώντας κάποιες δυνατότητες διείσδυσης βαλιστικές, αποκτώντας και πιο εξελιγμένους πυράβλους, ή μπορεί να το κάνει πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό πυράβλων που έχει, έτσι ώστε να πλημμυρίσει την αντιπυραυλική άμυνα ε, του αντίπαλου και να την καταστρέψει με τον τρόπο αυτό. Γι' αυτό η αντιπυραυλική άμυνα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόλυτη ασπίδα και με ένα όρο ασπής δεν με ικανοποιεί γιατί δημιουργεί κάποιες λανθασμένες εντυπώσεις. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση, από το ανακοινθέν που βγάλαμε στην Λισαβόνα. Δεν μπορεί να μιλάμε για ασπίδα που θα ασφαλίσει την Ευρώπη και θα κοστίσει μόνο 200 εκατομμύρια ευρώ. Ε, δεν υποτελεί πλήρη κάλυψη και γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχεί η Ρωσία. Όποιο σενάριο και να προκρίνουμε, μετά από 20 χρόνια για παράδειγμα ή ακόμα και πριν την εκπνοή της περίοδου αυτής, η Ρωσία θα μπορεί να ξεπεράσει αυτό το αντιρροπαϊκό σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ευκρινήσεις που δώσατε. Προηγουμένως εγώ αναφέρθηκα στο ευρωπαϊκό δυναμικό. Είπαμε ότι δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση. Συμφωνήσαμε λοιπόν με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Αμυντικής Βιομηχανίας και Εξοπλιστικής Βιομηχανίας να κάνουμε κάποια βήματα και θα ήθελα να καλέσω και τους επόμενους στο βήμα. Euh, euh, έχουμε λοιπόν την κυρία Σαμεγιάκ από την MBDA. Είναι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση κατασκευής ε, πυράβλων και έχουμε και τον στρατηγό κύριο Λιπάς από το Τάλις. Και σίγουρα αυτή η πρόσκληση μπορούσε να έχει απευθυνθεί και σε άλλους εκπροσώπους των ε, βιομηχανικών κύκλων την ADS αστριών που για παράδειγμα θα μπορούσε να μας βοηθήσει με τις απόψεις σας. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Έχει πιεστεί, συμπιεστεί μάλλον πολύ το δικό σας πάνελ. Σας παρακαλώ να προχωρήσετε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσω μιλώντας στα αγγλικά. Βεβαίως η προφορά μου είναι έντονα γαλλική, αλλά θα προσπαθήσω τουλάχιστον να πω δύο λόγια μόνο. Να σας εξηγήσω ακριβώς ποια είναι η MBDA. Είναι μια επιχείρηση που έχει ηγετικό ρόλο στον κόσμο για τα πυραυλικά συστήματα με εγκαταστάσεις στη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συστάθηκε το 2001. Αποτελεί τμήμα της ε, του συνδυασμού των εγκαταστάσεων των πυραυλικών που άνοικαν στην EADS, στην BAE Systems και στην Mechanica και συνδυάζει 50 χρόνια εμπειρία στα πυραυλικά συστήματα. Στόχος της παρουσίασής μου είναι να σας δώσω μια επισκόπηση αυτό, από το ποια θα μπορούσε να είναι η ευρωπαϊκή συμμετοχή ε, ε, στις αποστολές και στο δυναμικό ε, βαλιστικών πυράβλων της Ευρώπης για να δούμε ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε εμεί στην Ευρώπη, μπορούμε να πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα από διάφορε πλευρέ. Πρώτα απ' όλα, πλήρη ανάλυση τη βαλιστικής απειλής. Μία απειλή η οποία πολλαπλασιάζεται και να δούμε πού έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εκραγεί. Έτσι λοιπόν η ανάλυση που θα κάνουμε μας επιτρέπει να βρούμε το σωστότερο ε, σύστημα άμυνας. Η αμερικανική προσέγγιση ακολουθεί την ε, αρχή της στρατη... χάραξης στρατηγικής για το θέμα των βαλιστικών πυράβλων. Εμείς δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αγνοήσουμε τα όσα κάνουν οι Αμερικάνοι. Μπορούμε να δούμε λοιπόν και να ρωτήσουμε πώς η Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ε, με τρόπο που να συμπληρώνει τις δράσεις των ΗΠΑ. Και το τρίτο σημείο θα πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο για να χρησιμοποιήσουμε τα όσα έχουν ήδη γίνει στο παρελθόν και σε επίπεδο ε, βιομηχανικής κατασκευής αλλά και δυναμικού, ακολουθώντας μια σταδιακή προσέγγιση η οποία θα ελαχιστοποιήσει το κόστος. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αυτό ακούστηκε και προηγουμένως. Μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η Γαλλία και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε χρηματικό και σε τεχνικό επίπεδο, επαναλαμβάνω τι προσπάθειες των ΗΠΑ. Το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα είναι ο ορισμό της απειλής. Εδώ και πολλά χρόνια παρατηρούμε πως κάποια κράτη κάνουν συνεχείς προσπάθειες για να αποκτήσουν βαλιστικό οπλοστάσιο γιατί τέτοιου είδους οπλοσπάστιο αποτελεί την, ε, τις δυνάμεις των φτωχών. Έχουν χαρακτηριστεί έτσι. Οι χώρες αυτές θέλουν να γίνουν περιφερειακές δυνάμεις, αλλά δεν έχουν το, την απαραίτητη αεροπορία που θα τους επιτρέψει κάτι τέτοιο είτε γιατί για να αποκτήσει κανείς αεροπορική υπεροχή πρέπει να βρίσκεται σε συμμαχία, είτε γιατί χρειάζεται να αποκτήσεις επιθετικά αμήνα, ε, όπλα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, σε άλλους ελληνικούς αντί ε, για ε, αεροπορικές δυνάμεις με τον τρόπο που εμείς τις χαρακτηρίζουμε. Άρα λοιπόν, μπορούμε να δούμε ποια είναι η εμβέλεια. Πρέπει να είναι 3.000 ε, χιλιόμετρα και χωρί τη βοήθεια κάποιες πυρηνική δύναμη, τα κράτη αυτά δεν θα έχουν στη διαθέσή του την απαραίτητη τεχνολογία για να κατασκευάσουν ε, πυράβλους ε, τέτοιου ελληνικούς. Άρα λοιπόν, χωρίς την τεχνολογική βοήθεια από κάποια μεγάλη πυρηνική δύναμη, οι χώρες της διασποράς θα αποκτήσουν μόνο ε, βαλιστικούς πυράβλους μικρού και μέσου ελληνικούς, που θα τους δώσουν βέβαια το στάτους της περιφερειακής δύναμης, αλλά μόνο για την περιοχή τους. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και η ΕΠΑ θεωρούν πως οι μικρής και μέσης εμβέλειας βαλιστική πυραυλή αντιπροσωπεύουν το 93% του υφιστάμενου πυραυλικού οπλοστασίου, ενώ η απειλή για μεγάλου βεληνικούς ε, έχει εκτιμηθεί στο 6 μόνο Κατανοούμε λοιπόν πως για τις δυτικές χώρες η βαλιστική αυτή απειλή γίνεται πραγματική και πιθανή ε, στα ε, θέατρα επιχειρήσεων που είναι μακριά από τις χώρες μας. Έτσι λοιπόν οι χώρες διασποράς αποκτούν αυτή, αυτές τις βαλιστικούς πυράβλους για να καλύψουν τα δικά τους συμφέροντα και ε, κάνουν τα εξή τρία που είναι η βελτίωση της ακρίβειας, της επιχειρησιακής δυνατότητας ε, και του βεληνικούς. Όλες αυτές λοιπόν οι εξελίξεις μας δίνουν μία ιδέα για το τι θα συμβεί με, τις, με, βαλιστικές, με τους βαλιστικούς πυράβλους νέας γενιάς ε, που θα είναι πιο αποτελεσματικοί και θα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες διείσδυσης. Τι κάνουν οι ΙΠΑ. Η ΕΠΑ έχει ασχοληθεί με το θέμα και έχει δει και την πολιτική και την επιχειρησιακή και την βιομηχανική και την τεχνολογική διάσταση. Η νέα ε, προσέγγιση του ΝΥΠΑ παρουσιάστηκε από τη νέα διοίκηση σε τέσσερις φάσεις έτσι ώστε τα συστήματα άμυνας να προσαρμόζονται καλύτερα στις απειλές και γι' αυτό ε, στηρίζονται πιο πολύ από τις χώρες σημασίες ε, και από το ΝΑΤΟ. Ε, στη Σύνοδο της Λισαβόνας την περασμένη εβδομάδα αποφασίστηκε η επιχειρησιακή αεροπορική ασπίδα ή αν θέλετε άμυνα και οι ΕΕΠΑ ήδη έχουν αποφασίσει να συνεισφέρουν μέσω της σταδιακής προσαρμοστικής προσέγγισης που βασίζεται στα συστήματα SM3 Aegis για να αναχαιτίζουν στην έξω ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή περιμένουν την ευρωπαϊκή απόκριση. Το ΝΑΤΟ επίσης κάνει μία μελέτη για την βιομηχανική διάσταση του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ όπου ε, η έκθεση αυτή θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Επίσης, συστήνει να υπάρχει καλύτερη εναρμόνιση στην αμυντική βιομηχανία των συμμετεχόντων κρατών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία και η εμπλοκή αυτής αποφεύγουν στον διευρυνθεί το ε, τεχνολογικό κενό στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των δύο όχθων του Ατλαντικού. Αυτό που κάνουμε σήμερα λοιπόν στην Ευρώπη ε, και στις ευρωπαϊκές χώρες είναι το επόμενο κεφάλαιο που θα σας παρουσιάσω. Όπως ακούστηκε σήμερα το πολύ, η MBDA αλλά και άλλες εταιρείες έχουν ήδη εμπλακεί ε, σε δύο ε, είδη αντιαεροπορικών συστημάτων. Έχουμε πρώτα το Άστερ, και στην οικογένεια αυτών των όβλων με διαφορετικές χρήσεις, ε, είτε είναι εδάφους-εδάφους, είτε ε, η εκτόξευση γίνεται από πλοία και είναι ένα σύστημα το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ινωμένο Βασίλειο. Το σύστημα αυτό έχει σκοπό να επιτρέψει τα ευρωπαϊκά κράτη να επιτρέψουν, ε, να, προστατεύουν τα στρατεύματά τους εξωτερικά θέατρα μαχών και πρέπει να σας πω πως μέσα Οκτωβρίου πρόκειται ε, τα συστήματα αυτά, τα SMPT, να τα αξιολογήσουμε ε, για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν βαλιστικές απειλές. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις δοκιμές που έχουμε κάνει σε επιχειρησιακό περιβάλλον, η αναχέτηση ήταν επιτηλής. Έχουμε ακόμα και άλλη μία αντιεροπορική άμυνα, που είναι το σύστημα MIDS, το οποίο έχουν αναπτύξει ε, από κοινού η ΕΠΑ, ΕΕ, η Γερμανία και η Ιταλία. Όπου... Ο πλοίαρχος έχει το ραντάρ και τους εκτοξευτές, εκτοξευτήρες υπό τη διοίκηση και έλεγχό του. Έχουμε λοιπόν τα άλλα συστήματα και το Άστερ και το ΜΙΤ που θεωρούνται ως εθνικοί πόροι ε, που συνεισφέρονται στο πρόγραμμα ε, αντιπυραυλικής άμυνας ALTBMD του ΝΑΤΟ. Εφόσον οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποφασίσει να αναπτύξουν αυτά τα συστήματα, η απειλή βαλιστικών πυράβλων ε, άλλαξε γιατί έχουμε συνεχείς εξελίξεις και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πώς μπορούμε λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε, τι σύστημα ανώτερης ατμόσφαιρας μπορεί να αναπτυχθεί που να είναι και προσβάσιμο από τα κράτη της Ευρώπης. Το σύστημα που έχουμε που βασίζεται στα Aster System έχουν τη δυνατότητα να μεταλλαχθούν, έτσι ώστε να προστατεύσουν τις ενόπλες δυνάμεις ε, που έχουν αναπτυχθεί εναντίον των απειλών και που απειλούν να περιορίσουν τις πολιτικές και επιχειρησιακές τους δράσεις μέσω, για παράδειγμα, βαλιστικών πυράβλων. Ε, αυτό συμβαίνει ε, με τις βαλιστικούς πυράβλους μέσου και μικροβεληνικούς νέας γενιάς. Θα έχουμε όμως το νέο αναχαιτιστικό πύραυλο Aster Block 2 που θα, ε, θα ενταχθεί στο σύστημα Άστερ και θα μπορέσει να δώσει αυτό το έξτρα δυναμικό που, που χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε με τον τρόπο να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις μικρού και μέσου ελληνικούς και με πολύ καλές επιδόσεις εναντίον των πυράβλων κρούζ. Ποια είναι τα συμφέροντα και γιατί είναι ενδιαφέρον για μας να έχουμε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Πρέπει να σας πω πως η βαλιστική πύραυλη είναι πολύ βασικό χαρτί για τη βιομηχανία μας. Είναι στρατηγικό θέμα, είναι βιομηχανική πρόκληση. Γιατί, Γιατί οι επιδόσεις που πρέπει να έχουν τα συστήματα άμυνα το κόστος τους, τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, είναι στοιχεία κλειδιά έτσι ώστε να μπορούμε να λάβουμε ε, τις σωστές και τις ε, ε, χρονικά εμπρόθεσμες αποφάσεις. Η βαλιστική άμυνα είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο. Σε πολιτικό επίπεδο ε, σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς να προλάβουμε, να προδικάσουμε τι θα συμβεί στην Ευρώπη και βεβαίως ε, λόγω και του νέου χρονοδιαγράμματος που έχει επιβάλει η διοίκηση Ομπάμα με τις τέσσερις φάσεις της σταδιακής ενσωμάτωσης. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η δυνατότητα ανάπτυξης του συστήματος Άστερ, και για να πετύχουμε συμφωνήσαμε και συμφωνήσαμε μάλιστα με, τον, με το Τάλις έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Η πετυχημένη δοκιμή μεταξύ των βαλιστικών, εναντίον των βαλιστικών απειλών επιβεβαιώνουν ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολλά και πως το θάλις και σάφραν μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις των ε, όπλων αστέρ και όλα αυτά θα ενταχθούν σε ένα σύστημα παγκόσμιο διαλειτουργικό με το BMC3 του ΝΑΤΟ. Αυτά τα συστήματα που έχουν μειστοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν απειλές ε, στα ανώτερα και χαμηλότερα επίπεδα της ατμόσφαιρας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες ε, γενναίες βαλιστικών πυράβλων, για παράδειγμα τους ε, στόχους που μετακινούνται, θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με το SM3 και το TAD. Και μας δίνουν πολλά πλεονεκτήματα, δηλαδή αυξάνεται το επίπεδο συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ λόγω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, ενισχύουν το ρόλο ε, του BMC3 του ΝΑΤΟ, γιατί δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασία μεταξύ ε, Αμερικανών και Ευρωπαίων και βεβαίω ε, γίνεται μεγαλύτερη δέσμευση και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ συμμάχων. για να δικαιολογήσουμε τη συμμετοχή μας στην επιχειρησιακή δράση στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, γιατί όλα τα, θα πρέπει να διαπιστώσουμε πως τα όπλα που προτείνουμε είναι αμερικανικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει με κάποιο τρόπο το κενό αυτό να το καλύψουμε. Επίσης, έχουμε το, τα συστήματα ε, PAA των ε, Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία ε, θα πρέπει και εμείς να δημιουργήσουμε τα αντίστοιχά τους, έτσι ώστε να έχουμε αυτόνομη και προσαρμοσμένη στην ανάγκη μας άμυνα και να συνεργαστούμε με τις ΕΠΑ, οι ίσης όρους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως η συμμαχία θα είναι απόλυτα προστατευμένη από την βαλιστική απειλή. Σας ευχαριστώ. Για τους ανέχητιστές, να σας πω πως αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν, δύο λόγια για την εταιρεία Θαλής. Απασχολεί 60.000 άτομα. Έχει εγκαταστάσει σε 50 χώρες και στις περισσότερες ευρωπαϊκές. Η εταιρεία αυτή έχει μεγάλη εμπειρία, πάνω από 50 χρόνια, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των ραντάρ και των αμυντικών συστημάτων στον χώρο του διαστήματος, της αεροναυτιλίας, ε, όπως επίσης και στα χερσαία ε, συστήματα. Η εταιρεία μπορεί να χειριστεί όλες τις τεχνολογίες που έχουν σχέση με τους βαλιστικούς πυράβλους. Ξεκινώντας, θέλω να πω δύο λόγια για τα συστήματα ε, άμυνας βαλιστικών ε, πυράβλων από τεχνική καταρχήν άποψη. Από τεχνική άποψη χρειάζονται πολλές λειτουργίες για αυτά τα συστήματα, παρακολούθ, δυνατότητες παρακολούθησης εντοπισμού ε, μέσω του δορυφόρων ή άλλων συστημάτων, ε, δυνατότητες αναχέτησης σε διάφορα επίπεδα πυράβλων Ήδη το ακούσατε το θέμα από τη συναδερφό μου, ε, πύραυλη εν, ενδοατμοσφαιρική ή εξωατμοσφαιρική και επίσης όπως αναφέρθηκε σήμερα το πρωί δυνατότητες ελέγχου και διοίκησης. Αυτές οι δυνατότητες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πυραυλικής άμυνας. Τώρα, από τεχνική άποψη, η φιλοδοξία των συστημάτων ε, εξαρτάται από δύο θέματα. Το μέγεθος της περιφέρειας που θέλουμε να ε, ε, περιφρουρήσουμε και την, ε, το Βελινεκές. Τώρα, οι, τα δύο είδη άμυνα βασικά διαφέρουν λόγω αυτών των κριτηρίων. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια ευρύτερη περιοχή με μεγαλύτερες, μεγαλύτερο Βελινεκές των πυράβλων Αυτή είναι η εδαφική άμυνα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μικρότερο βεληνικές των εισερχομένων πυράβλων και ε, περιορισμένες περιοχές υποπροστασία. Αυτές, αυτή είναι η πυραυλική άμυνα θεάτρου, αλλά, ε, θεάτρου επιχειρήσεων. Ενδιάμεσα όμως ε, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες και κανείς δεν ξέρει ποια ποιο είναι το ακριβές όριο μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων. Φερρυπίν, στην Ευρώπη ενώ από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά η ευρωπαϊκή προσέγγιση θέλει να εγκαταστήσει ε, άμυνα για, από τους ε, πυράβλους θεάτρου επιχειρήσεων, η αμερικανική σκοπιά θέλει ε, άλλου είδους άμυνα. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο, κάποια συμπληρωματικότητα ε, με το θέμα της πυρηνικής αποτροπής. Ε, θέλω τώρα, όσον αφορά τις λεπτομέρειες, να αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Πρώτον, την απόφαση που έλαβε το ΝΑΤΟ για να αναπτύξει μια εδαφική πυραυλική άμυνα στην Ευρώπη ε, όπου πρέπει να εμπλακεί και η Ατλαντική ε, βιομηχανία. Δεν θα επανέλθω σε αυτά τα οποία αποφασίστηκαν στη διάσκεψη της Λισαβόνας, ανακούστηκαν σήμερα το πρωί. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι ρυθμίσεις ελέγχου και διοίκησης πρόκειται να αναπτυχθούν και να αποφασιστούν μέχρι τον επόμενο Μάρτιο, δηλαδή εξαιρετικά σύντομα, και το πρόγραμμα δράσης της ε, υλοποίηση αυτής της δυνατότητας πρέπει να έχει αποφασιστεί μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Άρα βιαζόμαστε για να είμαστε λοιπόν έτοιμοι γέρος, αλλά και για να εξασφαλίσουμε την πολιτική αποδοχή και την ε, μετέπειτα ε, επιτυχία της εδαφικής ε, πυραυλικής άμυνας πρέπει να εμπλακεί η διατλαντική ε, βιομηχανία, που σημαίνει ότι και οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές επιχειρήσεις και τεχνολογία να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτού του είδους την επένδυση. Μία κατάσταση όπου όλοι θα ωφεληθούν. Η απόφαση να στηριχθεί ε, η δαφική πυραυλική άμυνα στο πρόγραμμα LTLP είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από αυτή τη σκοπιά, δεδομένου ότι το ε, ALT-BMD πρόκειται να ε, παραδοθεί από τη διατλαντική βιομηχανία. Τώρα, δεν ε, υπάρχει ανάγκη να ξαναμελετηθεί το όλο σύστημα ή να ξανατεθεί σε δημοπρασία, αλλά πρέπει το σύστημα να παραδοθεί από τη διατλαντική ε, βιομηχανία με βάση τις, ε, την, την ισχύουσα προσέγγιση του LTBMD. Επίσης, η διατλαντική συνεργασία μπορεί να παραδώσει τους ε, αισθητήρε του δικτύου, δηλαδή και τους δορυφόρους και τα ραντάρ, που θα ε, είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστεί ότι τα αμερικανικά συστήματα ε, θα είναι προσβάσιμα από τη σκοπιά των C2 και της ε, ενσωμάτωσης των αισθητήρων από πλατφόρμες που θα έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη και το δεύτερο σημείο είναι αυτό που ε, θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά μπορεί να ρυθμιστούν. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ήδη συμμετέχει σε όλα τα πεδία της ε, άμυνας, ε, θεάτρου επιχειρήσεων και της εδαφικής, και της άμυνας σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο. Καταρχήν, η δορυφόροι έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να εντοπίσουν την εκτόξευση και να χαρακτηρίσουν τον τύπο του εισερχομένου πυράβλου. Η Γαλλία έχει με επιτυχία αναπτύξει μια τεχνολογία ε, που ονομάζεται Demonstrator. Ε, ανακοίνωσε στη Λισαβόνα ότι θα παράσχει στους ε, συμμάχους πληροφορίες από ένα έγκαιρης προειδοποίησης δορυφόρων μέχρι το 2020. Δεύτερον είναι τα ραντάρ, είναι δύο ειδών τα ραντάρ τα λεγόμενα έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλου βεληνικούς, ε, περίπου καλύπτουν 5-6 χιλιόμετρα, είναι υπεύθυνα της για την παρακολούθηση του ε, πυράβλου από τη στιγμή που εκτοξεύεται και ενημερώνουν τα εισερχόμενα ε, ραντάρ για την περίπου για τη θέση του εισερχομένου πυράβλου. Δεύτερον, είναι ραντάρ ενσωμάτωσης, εντοπισμού και στόχευσης και αναχέτησης. Οι διερμηνείς ζητούν συγγνώμη, οι εντολές από την υπηρεσία μας είναι να διακόψουμε την ε, εργασία μας τώρα για να μπορέσουμε να εργαστούμε και το, και το απόγευμα. Important technologic issues including algorithms, emission power, signal treatment, accuracy, discrimination of targets need to be mastered and exploited